Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Όπως είναι φανερό πλησιάζουν οι χριστουγεννιακές γιορτές, φαίνεται να είναι ισχνή παρουσία στην αίθουσα. Έχουμε ως προσκεκλημένους την κυρία Μαύρου και τον κύριο Λουκά. Ο κύριος Λουκάς είναι ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης και Δικαιοσύνης και η κυρία Μαύρου, Υπουργό Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα ήθελα να τους καλωσορίσω ιδιαίτερα για την παρουσίαση των ε, πεπραγμένων και των επιτευγμάτων της Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών στην Κύπρο για το τελευταίο λοιπόν εξάμεινο κατά το οποίο ίσχυσε την εκπεριτροπής Προεδρία η Κυπριακή Προεδρία και επίσης να μας ενημερώσουν για το Συμβούλιο της 6ης Δεκεμβρίου για τα δικαστικά και εσωτερικά θέματα. Θα έχουμε καταρχήν την παρουσίαση και μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση. Θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Μαύρου, εάν θέλει να λάβει πρώτη το λόγο, έχετε το λόγο. Καλημέρα σε όλους σας. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επίσης λαμβάνοντας τον λόγο εξ ονόματος του συναδέλφου μου, του Υπουργού Δικαιοσύνη και Δημόσιας τάξη. θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μας απευθύνατε και για τη θαυμάσια συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου της Κυπριακής Προεδρίας. Και θα συνεχίσω την παρέμβασή μου στα ελληνικά, μου το επιτρέπετε. Ε, κύριε Πρόεδρε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω το έργο της Κυπριακής Προεδρίας και της εξελίξεις στα σημαντικότερα θέματα που διαχειριστήκαμε τους τελευταίους έξι μήνες που αφορούν μέρος του τομέα των εσωτερικών υποθέσεων. Για τα υπόλοιπα θέματα του τομέα αυτού καθώς και για τα θέματα δικαιοσύνης θα σας μιλήσει στη συνέχεια ο συνάδελφος ε, Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης η πρόκληση για μια αποτελεσματική και αξιοπρεπή Προεδρία ήταν για μας ένα μεγάλο στίχημα, ιδιαίτερα δεδομένης της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και των πιέσεων στη ζώνη του ευρώ, αλλά και της υποεξέλιξη κρίσιμης κατάστασης στη Συρία. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαμε μια ειλικρινή και επικοδομητική συνεργασία και ένα συνεχή διάλογο σε όλους τους ε, τομείς ε, με αποτέλεσμα να καταφέρουμε να έχουμε ε, απτά αποτελέσματα προς όφελος όλων των πολιτών. Όπως ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής αυτής και τον περασμένο Ιούλιο, στόχος μας ήταν η ολοκλήρωση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου μέχρι το τέλος του 2012, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σας διαβεβαιώνω ότι εργαστήκαμε σκληρά για τον στόχο αυτό, παρά τις δυσκολίες, έχοντας πρωτίστως ως γνώμονα τη διασφάλιση της ποιότητας των νομοθετημάτων και των δικαιωμάτων όσων χρειάζονται διεθνή προστασία, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τυχόν καταχρήσεις. Ε, τι, πού βρισκόμαστε σήμερα. Έχει επιτευχθεί πολιτική συμφωνία ως προς την οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής και τον κανονισμό του Δουβλίνου. Σημειώθηκε, πιστεύω, σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ως προς την οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου. Μετά και τον τρίλογο που είχαμε ψες, ε, μπορώ να πω ότι ε, τα σημεία πάνω στα οποία θα χρειαστεί να ε, δουλέψουμε έχουν περιοριστεί σε ένα-δυο, αφορούν κυρίως τις ευάλωτες ομάδες. Το Συμβούλιο επίσης ενέκρινε τον Οκτώβριο του 2012 γενική προσέγγιση ως προς τον κανονισμό Eurodac, ο οποίος βασίζεται σε τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής της 30 Μαΐου του 2012. Δεδομένου ότι το Ευρωκοινοβούλιο ε, υιοθέτησε χτες μόλις τις ε, τροπολογίες του. Ε, ο πρώτος τρίλογος για το νομοθέτημα αυτό θα γίνει σήμερα. Θα ήθελα μόνο να παρατηρήσω ότι έχουμε φτάσει πολύ κοντά στην λήψη τελικών αποφάσεων για το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου είναι σημαντικό ε, όλες οι συνιστώσεις να κρατήσουμε και να αξιοποιήσουμε την δυναμική ε, που έχουμε πετύχει ώστε ο στόχος αυτός ε, να υλοποιηθεί σύντομα. Ε, στοχεύοντας σε ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου είναι ουσιώδες να επιδιώκουμε περισσότερες συγκλήσεις όχι μόνο νομοθετικές αλλά και πρακτικές. Είναι σημαντικό τα κρατη να έχουν στη διάθεση τους ουσιαστική υποστήριξη για να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Δηλαδή να υπάρχει συνεργασία και ειλικρινής και έμπραχτη αλληλεγγύη. Η Προεδρία παρακολούθησε στενά την εφαρμογή των συμπερασμάτων για το θέμα της αλληλεγγύης και στο Συμβούλιο ΔΕΗ στις αρχές του μήνα αυτού ενημέρωσε για την πρόοδο για τις δραστηριότητες που έχουν υλοποιηθεί ε, από τον Ιούνιο του 2012. Σε ό,τι αφορά την μετανάστευση, σημαντική πρόοδος επιτεύχθηκε στα υποσυζήτηση νομοθετήματα για τους εποχικά εργαζόμενους και τους ενδοεπιχειρησιακά μετατιθέμενους και είμαστε ήδη σε τριμερείς διαλόγους και για τα δύο αυτά ε, νομοθετήματα. Θα ήθελα να χαιρετήσω την έναρξη των τριλόγων μόλις ε, χθες για την οδηγία για τους εποχικά εργαζόμενους, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν στο επίπεδο του Συμβουλίου. Είμαστε σίγουροι ότι με την επικοδομητική συμβολή όλων τα νομοθετήματα αυτά δεν θα αργήσουν να οριστικοποιηθούν φέρνοντας μας ένα βήμα πιο κοντά σε μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική. Από μια τέτοια πολιτική δεν μπορεί να απουσιάζει το θέμα της ένταξης. Η διάσκεψη εμπειρογνωμόνων με θέμα το ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών που διοργανώθηκε τον Νοέμβριο ανέδειξε για ακόμη μια φορά την ένταξη ως κινητήριο μοχλό για ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή και ως κλειδί για τη μεγιστοποίηση των ωφελιών της μετανάστευσης. Επιπλέον, η Προεδρία εργάστηκε προς την αντιμετώπιση των προκλήσεων σε σχέση με την παράνομη μετανάστευση, με απόλυτο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Προς αυτή την κατεύθυνση παρακολουθήσαμε στενά την εφαρμογή της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μεταναστευτικές πιέσεις. Ιδιαίτερη σημασία δώσαμε και στον αγώνα κατά της εμπορίας προσώπων, που εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο υιοθέτησε τον Οκτώβρη συμπεράσματα σχετικά με τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλληψη της εμπορίας ανθρώπων. Επιπλέον, οργανώσαμε συνέδριο τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες για την περαιτέρω συνεργασία και συντονισμό ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για την πρόθεση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης ενάντια στην εμπορία προσώπων. Αναφέρω επίσης την δεύτερη έκθεση εφαρμογής του εγγράφου δράσης για την ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων που υποβλήθηκε στο ε, τελευταίο Συμβούλιο τώρα το Δεκέμβρη. Επίσης προωθήσαμε τις διαβουλεύσεις για την πρόταση του κανονισμού Eurosure. Με μεγάλη μας ικανοποίηση είχαμε χθε τον πρώτο τρίλογο για τον κανονισμό αυτό και επιβεβαιώσαμε την αμοιβαία ετοιμότητα για ειλικρινή και επικοδομητικό διάλογο με στόχο να τεθεί σε λειτουργία το Ευρωπαϊκό Σύστημα Παρακολούθησης Συνόρων κατά την προβλεπόμενη προθεσμία την 1η Οκτωβρίου του 2013. Πρόσθετα, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίηση της Προεδρίας για την επικοδομητική στάση του Ευρωκοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία μας επέτρεψε να καταλήξουμε σε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση για την πρόταση κανονισμού για τεχνικές τροποποιήσεις στον κώδικα ε, συνόρο Σέγγεν. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να έχει ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική αν δεν διατηρεί συνεχή συνεργασία και διάλογο με τις πιο σημαντικές χώρες προέλευσης και διέλευσης μεταναστών. Η Προεδρία επικεντρώθηκε ως εκ τούτου στην προώθηση της υλοποίησης των συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με την παγκόσμια προσέγγιση για τη μετανάστευση και την κινητικότητα. Έγιναν συγκεκριμένα και σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της σύναψης εταιρικών σχέσεων κινητικότητας με το Μαρόκο και την Τινησία, ε, ενώ με την Ιορδανία δρομολογήθηκε έναρξη διαλόγου που ελπίζουμε να οδηγήσει σταδιακά στη σύναψη εταιρικής σχέσης κινητικότητας. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σημαντικούς στρατηγικούς της εταίρους. Ε, με την Ινδία επιτεύχθηκε συμφωνία για τη θεσμοθέτηση συνεργασίας στη βάση μιας κοινή ατζέντα για την μετανάστευση και την κινητικότητα, ενώ με την Κίνα αποφασίστηκε η έναρξη ενισχυμένου διαλόγου και η πρόθεση σειρά συγκεκριμένων κοινών προγραμμάτων συνεργασίας. Ταυτόχρονα έχει συνεχιστεί και ενισχυθεί σημαντικά η συνεργασία μας με τη ΣΥΠΑ, με τις οποίες έχει συμφωνηθεί η υιοθέτηση ενός ανανεωμένου πλέον σχεδίου δράσης στα θέματα μετανάστευσης, ενώ με τη Ρωσία επίσης έχει εγκριθεί πρόγραμμα εργασίας που θα καλύπτει την ερχόμενη διετία. Θεμελιώδης αρχή της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης είναι το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης και των δικαιωμάτων που προκύπτουν από αυτή. Η Ένωση είναι κοινή αντίληψη ότι πρέπει να καταστεί πιο προσιτή για τους πολίτες της που πρέπει να είναι στο επίκεντρο όλων των πολιτικών, άρα πρέπει να είναι και ενήμερη για τις πολιτικές αυτές και για τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Προς αυτή την κατεύθυνση καταφέραμε σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σας ευχαριστώ γι' αυτό να ολοκληρώσουμε τις διαβουλεύσεις για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013 που είμαστε σίγουροι πως θα έχει ένα αξιόλογο και μακρόπνο αντίκτυπο στην προσπάθεια που καταβάλλεται για να φέρουμε την Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στους κανονισμούς που αφορούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία εσωτερικών υποθέσεων κάτω από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η συζήτηση των εν λόγω προτάσεων κανονισμών αποδείχθηκε πραγματική πρόκληση. Το θέμα αυτό ήταν από τα πιο δύσκολα και πολύπλοκα θέματα κατά την Προεδρία μας, ιδιαίτερα λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που επικρατεί ε, στην υπόλοιπη, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά είναι πραγματικά με ιδιαίτερη ικανοποίηση που αναφέρω ότι καταφέραμε να εξασφαλίσουμε μερική γενική προσέγγιση για τον οριζόντιο κανονισμό και τον κανονισμό για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας ε, Συνόρων και Θεωρήσεων. Ελπίζω αύριο στην Κορεπέρ να εξασφαλίσουμε συμφωνία για τον κανονισμό για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης και τον κανονισμό για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας αστυνομικής συνεργασίας. Ιδιαίτερα σημαντική θεωρούμε την προώθηση των δύο προτάσεων για αύξηση, αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης για την υλοποίηση προγραμμάτων solid για τα κράτη-μέλη που λόγω των σοβαρών συνεπειών της οικονομικής κρίσης έχουν δεχθεί βοήθεια από το μηχανισμό στήριξης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα αγαπητέ Πρόεδρε το Ευρωκοινοβούλιο για το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξε σε σχέση με την πρόθεση των δύο αυτών προτάσεων. Ολοκληρώνω την παρουσίασή μου λέγοντας ότι κατά την Προεδρία μας προσπαθήσαμε με ειλικρίνεια και αφοσίωση να ενεργήσουμε ως ένας έντιμος διαμεσολαβητής. Οι προσπάθειες μας επικεντρώθηκαν στο στόχο της δημιουργίας μιας καλύτερης Ευρώπης, στο πνεύμα των θεμελιωδών αρχών της Ένωσης που να σημαίνει περισσότερα για τους πολίτες της, με αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή προς μια Ευρώπη πιο κοντά στους γειτονές της. Είμαι σίγουρη πως και η επερχόμενη Ιρλανδική Προεδρία θα συνεχίσει τις κοινέ μας προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Σε κάθε προσπάθεια που κατέβαλε η Προεδρία η συμβολή του Ευρωκοινοβουλίου ήταν ε, πραγματικά ε, πολύτιμη και γι' αυτό οφείλω να εκφράσω ξανά τις θερμές μου ευχαριστίες. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Με το πέρας της τοποθέτησης του συναδέλφου Υπουργού θα είμαστε στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια είναι πιθανόν να έχετε. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. your turn, Mr. Luca. Ευχαριστώ κύριε Μαύρο. Κύριε Λουκά, η σειρά σα για να ολοκληρώσετε την παρουσίαση στον τομέα τη δικαιοσύνη. Κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για την ευκαιρία που μα δίνετε να παρουσιάσουμε το έργο που επιτέλεσε η Κυπριακή Προεδρία κατά το δεύτερο εξάμεινο του 2012. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, στον τομέα τη ασφάλεια και τη αστυνομική συνεργασία, η Κυπριακή Προεδρία έθεσε εξ αρχής ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση των προκλήσεων, πολλές εκ των οποίων εκ της φύσεώς τους, διασυνοριακές και διατομιακές, στοχεύοντας στην οικοδόμηση μιας ανοιχτής και ασφαλούς Ευρώπης μέσω της εφαρμογής της στρατηγικής εξωτερικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, η Κυπριακή Προεδρία έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση της αστυνομικής συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών με στόχο την καταπολέμηση του διασυνοριακού σοβαρού εγκλήματος, στην καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, περιλαμβανομένων των διαφόρων μορφών παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο, στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και τη διερεύνηση σχηματοοικονομικών συναλλαγών, στην εμπορία κλοπημένων έργων πολιτιστικής κληρονομιάς, και σε ό,τι αφορά την τρομοκρατία δόθηκε έμφαση στην περαιτέρω εφαρμογή των τεσσάρων πυλώνων της Ευρωπαϊκής Αντιτρομοκρατικής Στρατηγικής. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά θέματα τρομοκρατίας, η Κυπριακή Προεδρία προέκρινε την υιοθέτηση συμπρασμάτων Συμβουλίου αναφορικά με την προστασία ευάλωτων στόχων από τρομοκρατικές επιθέσεις. Τα συμπεράσματα αυτά καταδεικνύουν τη σημασία που πρέπει να δοθεί σε αυτόν τον τομέα, ιδιαίτερα μετά το πρόσφατο τρομοκρατικό χτύπημα στη Βουλγαρία και αποτελούν έναν πρώτο βήμα για περαιτέρω ενίσχυση των δημοσίων χώρων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διατηρώντας τους χώρους αυτούς ανοιχτούς με ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό. Περαιτέρω, η Προεδρία προώθησε την υιοθέτηση συμπερασμάτων Συμβουλίου αναφορικά με την ασφάλεια των αερομεταφορών από την τρομοκρατική απειλή, τα οποία εστιάζουν ιδιαίτερα στην επέκταση των δραστηριοτήτων αξιολόγησης κινδύνων στον τομέα της ασφάλειας των αεροπορικών μεταφορών. Θεωρούμε ότι η ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών παραμένει θέμα υψηλής προτεραιότητας και έτσι απότερος στόχος πρέπει να είναι η προστασία όλων των εμπλεκόμενων όπως οι επιβάτες και οι εργαζόμενοι στους αερολιμένες. Επιπρόσθετα, σε ό,τι αφορά θέματα τρομοκρατίας εκπονήθηκε έκθεση στην οποία καταγράφεται η πρόοδος που έχει επιτευχθεί αναφορικά με την εφαρμογή των συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την ενίσχυση των εσωτερικών και των εξωτερικών πτυχών του αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Περαιτέρω, η Προεδρία προέβηκε σε αναθεώρηση του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον τομέα της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης. Στον τομέα της ασφάλειας και της καταπολέμησης του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, η Κυπριακή Προεδρία έδωσε συνέχεια στο θέμα της λειτουργίας του Κέντρου Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, εξετάζοντας την εξωτερική διάσταση της εφαρμογής του προγράμματος. Σε κοινή συνεδρία της Επιτροπής ΚΟΖΗ με την, Επιτροπή, ε, με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης τον περασμένο Οκτώβριο συζητήθηκε ο σχεδιασμός με βάση τον οποίο η PSC θα λειτουργήσει ως σύνδεσμος ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας του κέντρου με τρίτες χώρες. Επιπρόσθετα, η Προεδρία προώθησε τη δημιουργία οριζόντιας ομάδας φίλων της Προεδρίας με στόχο την αναβάθμιση του συντονισμού στο επίπεδο του Συμβουλίου καθώς και την υποστήριξη της ανάπτυξης κοινή προσέγγισης και συνοχής σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Σε ό,τι αφορά την πάταξη του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματο και ειδικότερα όσον αφορά την ανάπτυξη ενό ευρωπαϊκού συστήματο μητρώων ονοματών επιβατών, το γνωστό PNR, θέλω να επισημάνω ότι το Συμβούλιο έχει πιστεί για την ανάγκη ύπαρξη τέτοιου συστήματο. Η ανάγκη αυτή καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική αν λάβουμε υπόψη ότι η Ένωση έχει ήδη συνάψει συμφωνίε με τρίτε χώρε οι οποίε επιτρέπουν την πρόσβαση ξένων υπηρεσιών σε δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών που ταξιδεύουν προ τι χώρε αυτέ. Αλλά δεν έχει ακόμη ρυθμίσει τη διαχείριση των θεμάτων αυτών από τι αρχέ των κρατών μελών σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπογραμμίζουμε το γεγονό ότι η απουσία κοινοτική ρύθμιση επί του θέματο αυτού δεν εμποδίζει τα κράτη-μέλη να εγκαθιδρύσουν το δικό του σύστημα PNR σε εθνικό επίπεδο, όπως έχουν άλλωστε ήδη πράξει ορισμένα άλλα κράτη-μέλη. Η θέσπιση μιας οδηγίας PNR ακόμα αφορά επιλογή μεταξύ της ρύθμισης της συλλογής και χρήσης δεδομένων επιβατών σε εθνικό επίπεδο ή της μη ρύθμισης του θέματος, οπότε θα επαφίεται στα κράτη-μέλη να πράττουν κατά το δοκούν. Το Συμβούλιο προσβλέπει με επικοδομητικό πνεύμα στη διαπραγμάτευση του κειμένου της οδηγίας με τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές. Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία PNR μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και του Καναδά, όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμη υποβάλει στο Συμβούλιο κείμενα προσχέδια τη συμφωνία. Καλούμε επί τούτο την Επιτροπή, όπως εντατικοποίηση τη διαπραγματεύσης και διαπραγματευτεί σκληρά, ούτω ώστε να έχουμε ένα κείμενο συμφωνία το συντομότερο δυνατό, παρόμοιο με αυτή παρόμοιο με αυτής με την Αυστραλία, ούτω ώστε να ικανοποιεί τα κράτη-μέλη και το Ευρωκοινοβούλιο. Στο πλαίσιο επίση τη πάταξη του οικονομικού οργανωμένου εγκλήματο, η Κυπριακή Προεδρία έχει προχωρήσει με την υιοθέτηση τη τελική έκθεση του 5ου γύρου αμοιβαίων αξιολογήσεων που αφορούσε ακριβώ το οικονομικό έγκλημα και διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση αυτή αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης κατά το Συμβούλιο ΔΕΗ τον Οκτώβριο. Το κείμενο της έκθεσης έτυχε ευρεία υποστήριξη ανάμεσα στους υπουργού και το έργο σε αυτόν τον τομέα θα συνεχιστεί με στόχο την περαιτέρω βελτίωση του νομοθετικού και του οργανωτικού πλαισίου σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση και την πρόληψη του οικονομικού εγκλήματο. Κατά τι συζητήσει, επισημάνθηκε στι αντιπροσωπείε των κρατών μελών η διαδικασία παρακολούθηση τη εφαρμογή των συστάσεων που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις εκάστου κράτους μέλους. Σε ό,τι αφορά την επιχειρησιακή διάσταση στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, η κύρια εστίαση τη κυπριακή Προεδρία ήταν στην εφαρμογή του κύκλου πολιτική για την καταπολέμηση του οργανωμένου και του σοβαρού διεθνού εγκλήματο. Ευθύ με την ανάληψη τη Προεδρία προχωρήσαμε σε αναθεώρηση και περαιτέρω βελτίωση του πλαισίου Impact ω πλατφόρμα πολυμερού συνεργασία και την εφαρμογή των πολιετών στρατηγικών σχεδιασμών και την υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων δράση, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορεί να γνωρίζουν καλύτερα το ρόλο και τις ευθύνες τους για την εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων δράσης του 2013. Παράλληλα, συνεχίσαμε την παρακολούθηση της υλοποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων δράσης για το 2012, το γενικότερο συμπέρασμα της οποίας είναι ότι ο κύκλος πολιτικής εφαρμόζεται ικανοποιητικά, όμως υπάρχουν αρκετά περιθώρια βελτίωσης, ιδίως όσον αφορά την συμμετοχή των κρατών μελών, τη χρηματοδότηση, την ενημέρωση σχετικά με τον κύκλο πολιτική σε εθνικό επίπεδο και τη συμμετοχή των εθνικών συντονιστών Impact. Η Επιτροπή ΚΟΖΗ επικύρωσε επίση τα 8 επιχειρησιακά σχέδια δράση για το 2013, η υλοποίηση των οποίων αρχίζει με τη νέα χρονιά. Τέλο, αξίζει να αναφερθεί ότι η Προεδρία συνέχισε τι προσπάθειε που έγιναν από προηγούμενε Προεδρίε για την περαιτέρω ανάπτυξη τη διοικητική εναλλακτική προσέγγιση για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο. Δεδομένου ότι η διοικητική προσέγγιση είναι ένα από τα οριζόντια ζητήματα, κοινά σε όλε τι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματο, στα πλαίσια του, τρέχον, του τρέχοντος πρώτου κύκλου, αρχέ Οκτωβρίου, έχουν καθοριστεί οι στόχοι του δικτύου σημείων επαφή, για του επόμενου 12 μήνε. Το δίκτυο θα υποβάλει σχετική έκθεση πρόοδου το Σεπτέμβριο του 2013. Περαιτέρω όσον αφορά ειδικά τα θέματα της αντιμετώπισης του φαινομένου της πλαστογραφίας ταξιδιωτικών γράφων και της διασυνοριακής τους διάστασης, η Κυπριακή Προεδρία έχει εισηγηθεί την πρόθεση της δημιουργίας ενός εναρμονισμένου εγχειριδίου για τον εντοπισμό κατάχρησης ταξιδιωτικών εγγράφων, στο οποίο θα καταγράφονται αναλυτικά οι διάφοροι εξειδικευμένοι μεθόδοι ελέγχου που πρέπει να διενεργούνται σε ένα ταξιδιωτικό έγγραφο για σκοπούς εντοπισμού απάτης επί των ταξιδιωτικών εγγράφων και ταυτότητας. Το εν λόγω εγχειρίδιο θα αποτελεί βοήθημα στο έργο των Ευρωπαϊκών Αρχών που ασκούν έλεγχο σε σύνορα και κατ' επέκταση θα συμβάλλει στην ασφάλεια των σύνορων, την καταπολέμηση τη λάθρομετανάστευση και γενικά του διασυνοριακού εγκλήματος. Σε ό,τι αφορά θέματα ανταλλαγή πληροφοριών και ενδυνάμωση τη αστυνομική συνεργασία, η Κυπριακή Προεδρία, κρίνοντα ότι το, η έγκαιρη πρόσβαση σε ακριβεί και επικυρωποιημένε πληροφορίε αποτελεί ουσιώδες στοιχείο τη συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολή του νόμου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, προήγησε σε αξιολόγηση και εφαρμογή του υφιστάμενου κεκτημένου. Τα αποτελέσματα τα οποία παρουσιάστηκαν στο Συμβούλιο ΔΕΗ το Δεκέμβριο θα αξιοποιηθούν στα πλαίσια των μελλοντικών συζητήσεων σε σχέση με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ανταλλαγής Πληροφοριών. Σε ό,τι αφορά την ενδυνάμωση της αστυνομικής εργασίας σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, η Κυπριακή Προεδρία προώθησε τη δημιουργία του άτυπου δικτύου εμπειρογνωμόνων EU CultNet, με υιοθέτηση σχετικού ψηφίσματο με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση τη εμπορία κλοπημαίων έργων πολιτιστική κληρονομιά. Στο πλαίσιο επίση τη προτεραιότητα για ενδυνάμωση τη αστυνομική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, η Κυπριακή Προεδρία διοργάνωσε δύο κοινέ αστυνομικέ επιχειρήσει, στι οποίε συμμετείχαν τα πλήστα κράτη-μέλη. Η πρώτη επιχείρηση, με την επωνομασία SICAR, στόχευε στον εντοπισμό όχημάτων που εξάγονται παράνομα και εγγράφονται σε άλλα κράτη-μέλη. Η επιχείρηση αυτή επικεντρώθηκε στην καταγραφή του modus operandi που ακολουθείται, καθώς και στις διαδρομές που ακολουθούνται για την εξαγωγή τους. Η δεύτερη επιχείρηση, με την ονομασία Αφροδίτη, στόχευε στην ανταλλαγή πληροφοριών για την εισδροή μεταναστών στο εσωτερικό των κρατών μελών σε σχέση με τις μεταναστευτικές πιέσεις τις κύριες οδούς διακίνησης παράνομων μεταναστών, τις χώρες τόχου της παράνομης μετανάστευσης, τις χώρες προέλευσης των μεταναστών, τα μέσα διακίνησή τους και τη χρήση πλαστών παραποιημένων ταξιδιωτικών εγγράφων. Ιδιαίτερη έμφαση επίσης δόθηκε σε θέματα βία στην οικογένεια, όπου εκπονήθηκε ευρωπαϊκό εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών αναφορικά με το ρόλο των αρχών επιβολής του νόμου, στην αντιμετώπιση του προβλήματος της φθοράς των υποθέσεων, δηλαδή του φαινομένου της παρέκκλησης, εκτροπής ή και αποτυχημένης διεκπαιρέωσής τους, στο πλαίσιο του ποινικού συστήματος το οποίο υιοθετήθηκε στην Ομάδα Εργασίας Επιβολής του Νόμου και θα κυκλοφορήσει στα κράτη-μέλη. Στον τομέα καταπολέμησης των ναρκωτικών, η Κυπριακή Προεδρία πέτυχε να υιοθετήσει την, υιοθέτηση της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα ναρκωτικά για τα έτη 2013 μέχρι 2020. Πιστεύουμε ότι η νέα αυτή στρατηγική, η οποία είναι ισορροπημένη και εκπονήθηκε με βάση απτά στοιχεία ως προς τη διάσταση του προβλήματος, ανταποκρίνεται εξίσου στις ανάγκες προσφοράς και ζήτησης ναρκωτικών ουσιών και διαχειρίζεται επιτυχώς τις υφιστάμενες προκλήσεις στον τομέα των ναρκωτικών, όπως είναι η εμφάνιση νέων ψυχοτρόπων ουσιών, η συνεχώ αυξανόμενη αριθμή θανάτων λόγω ναρκωτικών, η δυναμική των αγορών παράνομων ναρκωτικών ουσιών και η διάσταση των πρόδρομων ουσιών. Αναφορικά με τι δύο νομοθετικέ προτάσει που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση τη διακυβέρνηση του χώρου Σέγγεν και αφορούν την εγκαθίδρυση νέου μηχανισμού αξιολόγηση Σέγγεν και την τροποποίηση του κώδικα συνόρου Σέγγεν, ούτω ώστε να θεσμοθετηθούν νέοι κανόνε όσον αφορά την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα σε εξαιρετικέ περιπτώσει, η Κυπριακή Προεδρία παρέμεινε προσιλωμένη στην εργασία με το Ευρωκοινοβούλιο με στόχο την εξέβρεση μιας κοινά αποδεκτής βάσης προς επίλυση των, διαφόρων, των διαφορών μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου. Θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμηση μου για την προθυμία που επέδειξε το Ευρωκοινοβούλιο να εργαστεί μαζί μα προ αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα να εκφράσω επίση την ιδιαίτερη εκτίμησή μου προ την Επιτροπή ΛΥΠΕ και του δύο εισηγητέ τη, την κυρία Βέμπερ και τον κύριο Κοέλιο, για την όλη προσέγγιση του κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων αυτών, εργαζόμενοι όλοι σκληρά από τον, από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Πιστεύω πραγματικά ότι μετά τις συναντήσεις που είχαμε έχει επέλθει τέτοια σύγκληση θέσεων που μας επιτρέπει να θεωρούμε ότι μια συνολική συμφωνία επί των δύο προτάσεων είναι εφικτή κατά, την κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας. Όσον αφορά την διεύρυνση του χώρου Σέγγεν, η Κυπριακή Προεδρία ήλπιζε ότι το Συμβούλιο θα μπορούσε να εκδώσει την απόφαση που προβλέπει την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σέγγεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στη Ρουμανία, σύμφωνα με την εντολή που είχαμε λάβει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο. Προς τούτη την κατεύθυνση κατεβλήθησαν ιδιαίτερες προσπάθειες. Όμως, με τα λύπης αναφέρομαι ότι μετά από διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους, κατέστη σαφέ ότι το, όλο θέμα δεν μπορούσε να τεθεί στο Συμβούλιο προ λήψη απόφαση για διερεύνηση του χώρου Σέγγεν. Παρά τα αυτά, η Κυπριακή Προεδρία προέβηκε σε ενέργειε που θα διευκολύνουν τη λήψη τέτοια απόφαση από το Συμβούλιο με την πρώτη ευκαιρία, το συντομότερο δυνατό, περιλαμβανομένη τη επισκόπηση τη εφαρμογή των μέτρων που θα συμβάλλουν στην επιτυχή διερεύνηση του χώρου Σέγγεν τα οποία έχουν καθοριστεί κατόπιν τη σχετική εντολή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Επιπρόσθετα, η Κυπριακή Προεδρία εργάστηκε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη προ την κατεύθυνση τη ολοκλήρωση του συστήματο πληροφοριών Schengen δεύτερη γενιά, SIS-2. Επί τούτου, έγινε προετοιμασία επί όλων των πτυχών για την διενέργεια των τελικών δοκιμών με την και τη μετάβαση του συστήματος SIS-2 στο σύστημα SIS-2 η οποία είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί περί τα τέλη Μαρτίου του 2013. Το ζήτημα αυτό τέθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο στις 20 Νοεμβρίου 2012 κατόπιν κάποιων ενδείξεων αναφορικά με προβλήματα στο εθνικό σύστημα της Φιλανδίας τα οποία δυνατόν να καταστούσαν αδύνατη την τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Όμω σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά το Συμβούλιο ΔΕΗ Δεκεμβρίου, διεφάνηκε στην πορεία ότι έχει εξευρεθεί μια ενδιάμεση λύση η οποία θα επιτρέψει την συμμόρφωση στο αρχικό χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λειτουργία του ΣΥΣ2, δηλαδή τον Μάρτιο του 2013. Σε ό,τι αφορά την υφιστάμενη διαδικασία αξιολόγηση τη ορθή εφαρμογή του κεκτημένου Σέγγεν, επιθυμώ να αναφέρω ότι η Κυπριακή Προεδρία ολοκλήρωσε και τι νέε αποστολέ που περιλαμβάνεται στο ημερολόγιο αξιολογήσεων για το έτος 2013. Επίσης, ετοίμασε και υιοθέτησε το ημερολόγιο αποστολών αξιολογήσεων για το έτος 2013. Συγγνώμη, προηγουμένως του 2012 και ετοίμασε και υιοθέτησε το ημερολόγιο αποστολών αξιολογήσεων για το έτος 2013. Στον τομέα του ποινικού δικαίου, η Προεδρία έχει εργαστεί σκληρά και πέτυχε γενική προσέγγιση στο Συμβούλιο ΔΕΗ Δεκεμβρίου αναφορικά με την πρόταση οδηγία, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση τη ικανότητα των κρατών μελών να δεσμεύουν και να δημεύουν προϊόντα εγκληματικών πράξεων. Η πρόταση αυτή, η οποία αποτέλεσε εξ αρχή μια εκ των προτεραιοτήτων τη Κυπριακή Προεδρία στον τομέα του ποινικού δικαίου, στοχεύει στη διασφάλιση πιο αποτελεσματικών μέτρων, μεθόδων, καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και στην ενίσχυση της συνεργασίας των αρμοδίων υπηρεσιών των κρατών μελών στον τομέα αυτό. Οι σημαντικότερες πρόνοιες της συμβιβαστικής προσέγγισης που έχει επιτευχθεί είναι συντομία οι ακόλουθες. Το πηδείο εφαρμογή της οδηγίας καλύπτει μόνο τα δικήματα που καθορίζονται στο άρθρο 88 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα λεγόμενα Eurocrimes εκτεταμένε εξουσίε δέσμευση περιορίζονται στα σοβαρά ποινικά δικήματα, τα οποία άμεσα ή έμεσα δημιουργούν παράνομο οικονομικό όφελο, σύμφωνα με την πολιτική καθοδήγηση των Υπουργών στο Συμβούλιο Οκτωβρίου ΔΕΗ Οκτωβρίου 2012. Η δίμευση χωρί καταδίκη περιορίζεται σε δύο μόνο περιπτώσει: τη μόνιμη ασθένεια και τη διαφυγή του υπόπτου ή κατηγορουμένου, παρέχοντας τη δυνατότητα εφαρμογή προνοιών εσωτερικού δικαίου για καταδίκη ερήμη. Η δέσμευση μπορεί να γίνει από αρμόδια αρχή πέραν από δικαστική αρχή σύμφωνα με το σύστημα που ισχύει σε ορισμένα χώρε κρατημέλη, νοουμένου ότι θα επιβεβαιωθεί το μέτρο από δικαστήριο ή δικαστική αρχή. Επίσης, προβλέπεται η λήψη μέτρων για δέσμευση ω επίγον μέτρων πριν από την έκδοση κανονικού διατάγματος δίμευση. Οι διασφαλίσει είναι λεπτομερεί και σε μεγάλο βαθμό όπως η αρχική πρόταση τη επιτροπή. Για τη διαμόρφωση του συμβιβαστικού κειμένου καθοδηγηθήκαμε από την ανάγκη διασφάλισης της αρχής της αναλογικότητας και σεφασμού των εχέγγυων που κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ορισμένα κράτη-μέλη επιθυμούσαν κάποιε πρόνοιε να είναι πιο φιλόδοξε, όπω για παράδειγμα αυτή τη δίμευση χωρί προηγούμενη καταδίκη. Το κείμενο που συμφωνήθηκε αποτελεί του ελάχιστου κανόνε και είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού. Επιτρέπεται στα κράτη-μέλη βεβαίω να προχωρήσουν πέραν από τι συγκεκριμένε πρόνοιε. Γενική προσέγγιση επιτεύχθηκε επίση το Συμβούλιο 2 Δεκεμβρίου και επί τη πρόταση οδηγία σχετικά με τι πράξει προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικέ πληροφορίε και τι πράξει χειραγώγηση τη αγορά, γνωστόν ω ΜΑΤ, η οποία έχει σκοπό την αποτροπή χειραγώγηση τη αγορά και κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω αποτελεσματικών ποινικών κυρώσεων. Το ΜΑΤ είναι ένα μέσο το οποίο προβλέπει ποινικέ κυρώσει και είναι συμπληρωματικό ως προς τον κανονισμό ΜΑΡ, ο οποίος προβλέπει την επιβολή διηγητικών κυρώσεων. Τα δύο αυτά νομοθετήματα αποτελούν μέρος του πακέτου προτάσεων μαζί με, τον, με την ΜΥΦΙΤ και την ΜΥΦΙΡ. Σημειώνεται ότι στις 5 Δεκεμβρίου 2012 επιτεύχθηκε Συμφωνία Γενικής Προσέγγισης και σε σχέση με το ΜΑΡ, η Προεδρία είναι τη άποψη ότι η γενική προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο τελευταίο Συμβούλιο ΔΕΗ αποτελεί μια καλή βάση για την έναξη των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο προέβησε ψηφοφορία προσανατολισμού όσον αφορά το ΜΑΡ και το ΜΑΤ στι 9 Οκτωβρίου του 2012. Επιπλέον, επί Κυπριακής Προεδρίας κατατέθηκε πρόταση οδηγίας για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμέσου του ποινικού δικαίου, PIF, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο εκτενώς συζητήσεων. Κατά τις συζητήσεις αυτής, αυτές αναδείχθηκαν πολύπλοκα ζητήματα τα οποία χρήζουν περαιτέρω μελέτης. Όσον αφορά την πρόταση για την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνα σε ποινικέ υποθέσει, με πρωτοβουλία τη Προεδρία επανήρχησαν οι για το θέμα και τον Οκτώβριο πραγματοποιήθηκε ένα τρίλογο ενώ ένας δεύτερος προγραμματισμένος τρίλογος ακυρώθηκε. Η Προεδρία συναντήθηκε με τα περισσότερα πολιτικά κόμματα του Ευρωκοινοβουλίου και εξήγησε τη θέση του Συμβουλίου καθώς και την ανάγκη υιοθέτηση αυτής της οδηγίας. Αναφορικά με την πρόταση οδηγίας για το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο, η Κυπριακή Προεδρία έχει επενδύσει πολύ χρόνο και ενέργεια. Παρά την πολύ επικοδομητική συνεργασία με τα κράτη-μέλη και τις καλές επαφές με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποδείχθηκε αδύνατο να επιτευχθεί συμφωνία σε αυτό το στάδιο, καθώ το Κοινοβούλιο απαιτεί περισσότερο χρόνο για να μελετήσει το φάκελο και να διατυπώσει τι θέσει του. Είμαστε βέβαιοι, ωστόσο, ότι το έργο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα είναι μια καλή βάση για την επίταξη συμφωνία στο εγγύ μέλλον. Σε ό,τι αφορά το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο στον τομέα τη δικαιοσύνη, το Συμβούλιο ΔΕΗ πέτυχε γενική, μερική γενική προσέγγιση επί των δύο προτάσεων για τη θέσπιση του κανονισμού δικαιοσύνη και του κανονισμού δικαιώματα, ισότητα και ηθαγένεια τον Ιούνιο του 2012. Η μερική γενική προσέγγιση κάλυπτε όλο το κείμενο των δύο κανονισμών με εξαίρεση δύο ζητήματα. Πρώτο, τα ποσά του προπλογισμού και δεύτερον το ερώτημα εάν μερικές πτυχές της πολιτικής περί ναρκωτικών θα πρέπει να καλύπτονται από το πρόγραμμα δικαιοσύνη. Όσον αφορά τα ποσά του προπλογισμού, για αυτά θα υπάρξει διαπραγμάτευση σε οριζόντιο επίπεδο σχετικά με τα ναρκωτικά. Η Προεδρία βρίσκεται στο το διάστημα αυτό σε συζητήσεις για να λύσει το πρόβλημα αυτό και είναι αποφασισμένη να βρει μια λύση μέχρι το τέλος του χρόνου. Τόσο το Συμβούλιο όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζουν την σημαντικότητα της κατάληξης σε συμφωνία επί των δύο κανονισμών. Σκοπός του προγράμματος δικαιοσύνη είναι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης όπου μέσω της δικαστικής συνεργασίας θα προωθείται η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, η κατάρτιση των δικαστών καθώς και του δικαστικού προσωπικού. Παράλληλα, το πρόγραμμα Δικαιώματα Ισότητα και στοχεύει στη δημιουργία ενός πλαισίου το οποίο θα προωθεί και ενισχύει ανάμεσα σε άλλα την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πρόληψη και καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και την προστασία των παιδιών. Ενέκα της εξαίρετης συνεργασίας μεταξύ του Ευρωκοινοβουλίου και της Κυπριακής Προεδρίας, οι τρίλογοι ξεκίνησαν άμεσα, αμέσως μετά την ψηφοφορία προς Ανατολισμού της 27 Νοεμβρίου 2012 και κατά τους τριλόγους αυτούς σημειώθηκε σημαντική πρόοδος. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν δύο τρίλογοι και από των δύο προτάσεων και έχει επέλθει συμφωνία σε σωρία ζητημάτων. Όσον αφορά το θέμα της προσχώρησης της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θα ήθελα να επισημάνω ότι το θέμα τέθηκε στην ημερησία διάταξη του Συμβουλίου ΔΕΗ Δεκεμβρίου. Οι διαπραγματεύσει έχουν επαναρχίσει και έχουν λάβει χώρα τρει γύρι διαπραγματεύσεων μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των άλλων κρατών μελών του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Δύο επιπλέον γύρι έχουν προγραμματιστεί για το 2013. Η Κυπριακή Προεδρία έχει επικεντρωθεί σε δύο παράλληλες οδούς Πρώτον, στα περιθώρια της ομάδας εργασίας για τα θεμελιώδη δικαιώματα, ΦΡΕΜΠ, e ως της ειδική Συμβουλευτικής Επιτροπής που προετοιμάζει τις διαπραγματεύσεις στο Στρασβούργο, ώστε να δίδεται συνεισφορά στον διαπραγματευτή της Ένωσης για τις διαπραγματεύσεις και δεύτερον, έχουμε εργαστεί εντατικά εππεριορισμένων στοιχείων των μελλοντικών εσωτερικών κανόνων που πρέπει να ετοιμαστούν στο πεδίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όσον αφορά το πακέτο των προτάσεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, που η Προεδρία είχε θέσει ως μία από τις βασικές προτεραιότητες της, προγραμματίστηκαν μέχρι σήμερα πέντε διήμερες συναντήσεις για τη συζήτησή τους και στις 19-20 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ακόμη μια συνάντηση που θα αφιερωθεί αποκλειστικά στην οδηγία. Στην πρόταση κανονισμού επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος στην κατάρθρωση συζήτησή του και κάλυψε και μέρος του κεφαλαίου 5, οριζόντια θέματα που, που απασχολούσαν τα κράτη-μέλη, όπως ο μεγάλος αριθμός των κατεξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων, το διοικητικό κόστος και η εφαρμογή κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων στο δημόσιο τομέα. Συζητήθηκαν τόσο στα πλαίσια της ομάδας TAPIX, όσο και στα πλαίσια της ομάδας φίλων της Προεδρίας που ενεργοποιήθηκε για το σκοπό αυτό. Θεωρούμε ότι έχει καταγραφεί πολύ σημαντική πρόοδος επί των ζητημάτων αυτών και έχουν αποσαφινιστεί πολλά θέματα. Ωστόσο, από τις συγκεκριμένες συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο διαπιστώθηκε ότι τα τρία ζητήματα δεν είναι απολύτως όρημα για τη λήψη απόφασης στο παροστάδιο. Για τον αριθμό κατεξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων, τα κράτη-μέλη συμφώνησαν ότι αυτός πρέπει να μειωθεί σημαντικά. Παρόλο που η Επιτροπή φάνηκε έτοιμη να προτείνει δραστική μείωσή τους, αυτό δεν ήταν τεχνικά εφικτό πριν ολοκληρωθεί η πρώτη ανάγνωση και συζητηθούν οι εναλλακτικέ λύσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αντί αυτών των πράξεων. Για το θέμα του διοικητικού κόστου, τα κράτη-μέλη συμφώνησαν ότι το μικρομεσαίο μέγεθο μια επιχείρηση δεν μπορεί να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για την εξαίρεσή της από τις υποχρεώσεις που προνοεί ο κανονισμός και φάνηκε να προτιμούν τη θέσπιση εξαιρέσεων με βάση την επικινδυνότητα που περιέχει η φύση των εργασιών της επιχείρησης και η επεξεργασία των δεδομένων. Για το θέμα του δημόσιου τομέα καταγράφηκαν οι ανησυχίε των κρατών μελών και συμφωνήθηκε ότι αυτό θα πρέπει να εξεταστεί ξανά μετά το πέρας της πρώτης ανάγνωσης από τα κράτη-μέλη όπου τα κράτη-μέλη θα έχουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το βαθμό ελαστικότητας που μπορεί να έχει. Πιο πάνω προσεγγίσεις των κρατών μελών και για τα τρία οριζόντια θέματα υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο ΔΕΗ που πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Δεκεμβρίου. Συγκεκριμένα συμφωνήθηκε όπως για το πρώτο ζήτημα που αφορούσε τη διαγραφή αρμοδιοτήτων και κατεξοδότηση πράξης και εκτελεστικές πράξεις και της αντικατάστασης τους με εναλλακτικέ προτάσεις, αυτό θα αποφασιστεί μετά την ολοκλήρωση της πρώτης επεξεργασίας του κειμένου του σχεδίου κανονισμού. Για το δεύτερο ζήτημα, για τις διοικητικές επιβαρύνσεις, το Συμβούλιο έχει δώσει εντολή στην Ομάδα Ανταλλαγή Πληροφοριών και Προστασία Δεδομένων, DAPIX, να συνεχίσει τις εργασίες τη επί συγκεκριμένων προτάσεων με σκοπό να εισαχθεί στο κείμενο του σχεδίου κανονισμού ενισχυμένη προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο. Και το τρίτο ζήτημα σχετικά με το κατά πόσον και με ποιον τρόπο ο κανονισμό μπορεί να εξασφαλίσει ευελιξία στο δημόσιο τομέα των κρατών μελών, αυτό θα αποφασιστεί μετά την ολοκλήρωση τη πρώτη εξέταση του κειμένου του σχεδίου κανονισμού. Όσον αφορά την πρόταση οδηγία, η Προεδρία προχώρησε στην κατάρθρον συζήτησή τη, ενώ όπω ανέφερα, εκκρίνει ακόμη μια συνάντηση. Με βάση τη συνθήκη τη Λισαβόνα, οι κανόνε προστασία προσωπικών δεδομένων πρέπει να τη χάνουν ομοιόμορφης εφαρμογή σε όλους τους πρώην πυλώνες της Ένωσης. Για να κάνω κάποια Βλέπω ότι ολοκληρώνεται σιγά σιγά. Αλλά αν μπορείτε κάπως να συνοψίσετε για να έχουμε και λίγο χρόνο για τη συζήτηση. Να αναφέρω ότι όσον αφορά την πρόταση της Βουλευτής με τη σχετικά με θέσπιση πολιετούς προγράμματος ε, πλαισίου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ΦΡΑ, η Προεδρία ε, ευχαριστεί την Επιτροπή ΛΥΠΕ για την επικοδομητική της στάση και την προθυμία σας να επιτευχθεί μια ισορροπημένη συμβαστική λύση σχετικά με το νέο πολιετές πρόγραμμα πλαισίου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Για, και ως εκ τούτου ε, η, η Προεδρία στα πλαίσια να βοηθήσει τον οργανισμό ΦΡΑ να μπορέσει να λειτουργήσει για το 2013 ε, προχώρησε και ενημέρωσε τον οργανισμό ότι μπορεί να συνεχίσει τις εργασίες του βάσει του, προγράμ, του τρέχοντος προγράμματος. Η λύση αυτή, αν και δεν είναι ιδανική, ε, ε, εμφανίζεται ως ο μόνος ρεαλιστικός τρόπος για να διασφαλιστεί ότι ο οργανισμός θα είναι σε θέση να συνεχίσει να εργάζεται χωρίς διακοπή. Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τόσο στον Πρόεδρο, όσο και στα μέλη της Επιτροπής ΛΥΠΕ, την ιδιαίτερη εκτίμηση και τις ευχαριστίες μου για την άψογη συνεργασία που είχαμε κατά το εξάμεινο που μας πέρασε για επίτευξη του κοινού στόχου της περαιτέρω εδραίωσης ενός χώρου δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you. Thank you both, Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μαύρο, ευχαριστώ κύριε Λουκά. Σας ευχαριστώ για τη λεπτομερή σας ε, παρουσιάση ε, και σας ευχαριστούμε που ε, αναγνωρίσατε την ετοιμότητα των μελών της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ στα πλαίσια της συνεργασίας με την Προεδρία σας. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους για τη συζήτηση. Προσπαθώ να δω ποιος έχει ζητήσει το λόγο. Έχουμε κάποιους κύριους βουλευτές εδώ. Βλέπω ότι η κυρία Ρομέρο Λόπες. Θέλετε να ξεκινήσετε, κύριε Ρομέρο. Ευχαριστώ. Πρώτο. το λόγο τόσο γρήγορα. Θέλω να... να... Θέλω να κάνω κάποιες παρεμβάσεις ε, για το σχόλιο των Υπουργών. Για την κυρία Μαύρου, καταρχήν, ε, για... Μάλλον, ε, να σας πω ότι για το πακέτο ασύλου εμείς ε, δεν είχαμε την ε, ίδια άποψη σε σχέση με το πώς συζητήθηκε το ζήτημα και δεν νομίζω ότι τώρα θα δούμε και την πραγματική συνεργασία στην οποία αναφερθήκατε γιατί το σύστημα του Δουβλίνου είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο δεν επιλύει τα προβλήματα για το μέλλον και πρώτος οδηγίας για τη Eurodac που εγκρίναμε χτες όλους ε, όσους ζητούν άσυλο τους μετατρέψαμε σε πλέον ευάλωτους. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που πρέπει να συζητηθούν ακόμη. Δυστυχώς δεν σημειώθηκε ένα βήμα προς τα μπρος με αυτό το πακέτο ασύλου. Δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν πάρα πολλά σημεία εκκρεμή και σε ό,τι αφορά τώρα για την πολιτική μετανάστευση, το ίδιο θα μπορούσα να σας πω, αλλά θα ήθελα καταρχήν να μου απαντήσετε για τις συμφωνίες που, έγιναν με το Μαρόκο και την Τινησία για το θέμα της κινητικότητας και πού μπορούμε να βρούμε τη σχετική τεκμηρίωση για τις ε, συμφωνίες που ανακοινώσατε με την Ινδία, με τη Ρωσία. Δηλαδή για όλες αυτές τις συμφωνίες τις οποίες αναφερθήκατε ότι μονογραφήθηκαν τώρα να στραφώ στον κύριο Λουκά για τον... Σα άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά καθ' όλη την παρέμβασή σα, αλλά τελικά δεν αναφερθήκατε στην οδηγία προστασία των δεδομένων, που όπως ξέρετε είναι ένα από τα θεμελιώδη και ουσιαστικά ζητήματα. Αγωνιστήκαμε πάρα πολύ για να γίνει η εξέταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παράλληλα με την εξέταση του κανονισμού, όμως δεν ακούσαμε τίποτα για την οδηγία αυτή. Τίποτα δεν μας είπατε. Και όπως ξέρετε αυτή η οδηγία αποτελεί το πλαίσιο βάσει του οποίου θα θεσπιστεί αυτή η προστασία των δεδομένων. Η προστασία των φυσικών προσώπων που στην πραγματικότητα πέρα από την προστασία ε, των ε, φυσικών προσώπων τελικά μιλάμε για έλλειψη προστασία των φυσικών προσώπων, ε, γιατί μιλάμε για κάποιε κατεξαίρεση περιπτώσει όπου θα πρέπει να παρέμβουν οι χώρε για να υπάρχει καλύτερη αστυνομική και δικαστική συνεργασία. Όμω βέβαια εσεί τίποτα δεν μα είπατε γι' αυτό, γι' αυτό ήθελα να σα ρωτήσω. Γιατί αυτή η οδηγία έχει μπλοκαριστεί, γιατί δεν προχωρά και γιατί δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στο πλαίσιο αυτό και ουσιαστικά αποτελεί τη βάση συζήτηση για πολλές άλλες εκκρεμείς προτάσεις ε, και αποπαιτούν συζήτηση όπως παίρνουμε το σχάρι τα PNR. Ο κατάλογος με τα ονόματα των επιβατών. Και θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω σε σχέση με τις δικονομικές εγγύσεις. Και αυτό το θέμα είναι εκρεμές. Αυτό το πακέτο δικονομικών εγγύσεων μιλήσατε για την δωρεάν νομική συνδρομή. Γιατί η Ευρώπη, όπως γνωρίζετε, και τώρα Συζητούμε σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΕΣΔΑ και όπως ξέρετε η δωρεάν νομική συνδρομή αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό δικαίωμα ε, ουσιαστικά βρίσκεται στον ε, ίδιο πυλώνα με το δικαίωμα χορήγησης αρρωγής ε, κατά την υποδοχή και ουσιαστικά τελικά γιατί μιλάμε ότι θα έχουμε ένα πακέτο δικονομικών εγγύσεων μόνο για τους πλούσιους, για αυτούς που έχουν χρήματα. Και εν τέλει δεν είναι αυτός ο πραγματικός τρόπος να αγωνιστούμε για την προστασία των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων για να είναι πραγματικότητα ο σεβασμός ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να καταπολεμήσουμε τον ρατσισμό, την ξενοφοβία κτλ. Αυτά είναι σημεία που όπου δυστυχώς δεν σημειώθηκε πρόοδος. Θα ήθελα να θέσω και άλλες ερωτήσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι μακρηγορήσατε και μου είναι αρκετά δύσκολο να συνεχίσω, γιατί θα ήθελα να αφήσω χρόνο και για τους υπόλοιπους. Όμως, μια τελευταία ερώτηση. Για το πρόγραμμα Αφροδίτη, το οποίο αναφερθήκατε σε σχέση με την είσοδο των μεταναστών, τι οδού, τι χώρε προέλευση κτλ. Μπορείτε να μα πείτε κάποιε λεπτομέρειε γι' αυτό. Το Συμβούλιο αποφάσισε επί αυτών των πτυχών και γιατί δεν υπάρχει ε, κάποια δράση, ανάληψη δράση σε σχέση με τις χώρες προέλευσης, δηλαδή να ξέρουμε από πού προέρχονται αυτές οι μεταναστευτικές ροές και αν, υπάρξει, αν έχει υπάρξει κάποια συνεργασία σε σχέση με αυτές τις χώρες, να μας ενημερώσετε σχετικά. Ευχαριστώ κύριος Παπα-Νικολάου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θέλω να ευχαριστήσω την Κυπριακή Προεδρία για την πολύ επικοδομητική συμβολή της στα θέματα τη δική μα επιτροπή το εξάμεινο που πέρασε. Γνωρίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, μια δύσκολη περίοδο για την Κύπρο, μια δύσκολη περίοδο για την Ευρώπη και βεβαίω μια κρίσιμη περίοδο για τα θέματα που πραγματευόμαστε σε αυτή την Επιτροπή, το πακέτο ασύλου, το, ζήτημα του Σέγγεν και, και πολλά από όσα αναφερθήκατε. Και νομίζω ότι μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες η Κυπριακή Προεδρία κατόρθωσε να, με συνέπεια να συμβάλλει επικοδομητικά στην πρόοδο των θεμάτων. Είναι δεδομένο ότι σε ένα εξάμεινο δεν είναι εφικτό να έχουμε ε, τελικά αποτελέσματα στα πάντα. Ε, γνωρίζω όμως ότι πολλές φορές μέχρι αργά το βράδυ ε, οι εκπρόσωποι της Προεδρίας βρισκόντουσαν σε συναντήσεις και σε διαπραγματεύσεις με μας, με την Κομισιόν. Ε, όλο αυτό το διάστημα, ε, παρά τα προβλήματα, την Κυπριακή Προεδρία την είχαμε κοντά μας και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να το καταδείξουμε. Μια μικρή χώρα συντέλεσε αποφασιστικά την περίοδο αυτή με την Προεδρία της στο να έχουμε πρόοδο σε πολλά θέματα. Ε, γνωρίζω ότι σήμερα στον απολογισμό είναι δύσκολο να αναφερθούμε έτσι με λεπτομέρειες σε πολλές πτυχές των θεμάτων. Η κυρία Λόπεζ ήδη έχει ερωτήσει πολλά. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση ε, σε σχέση με τη συνεργασία της Ευρώπης με τις τρίτες χώρες. Το προηγούμενο, το, προηγούμενο διάστημα είχαμε την Αραβική Άνοιξη, τώρα έχουμε τις εξελίξεις στη Συρία ε, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όλοι ότι για να μπορέσουμε να έχουμε μια αποτελεσματική πολιτική στο άσυλο, μια αποτελεσματική πολιτική μεταναστευτική, με αλληλεγγύη και κατανομή των βαρών, βασική προϋπόθεση είναι να μπορούμε να έχουμε ε, καλή συνεργασία και τη συνδρομή των τρίτων χωρών και σε ό,τι αφορά την επανεισδοχή των υπηκών τους και σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των χωρών αυτών προκειμένου να περιορίζουμε εν τη γενέση τους τις όποιες μεταναστευτικές ροές. Μέσα από την Προεδρία αυτό το εξάμεινο αισθάνεστε ότι έχουμε κάποια πρόοδο και δεν αναφέρομαι μόνο στην Τουρκία, αναφέρομαι ευρύτερα στις γειτονικές τρίτες χώρες και ευρύτερα σε σχέση με τα προβλήματα και την ε, ένταση που υπάρχει στη γειτονιά μας. Νομίζετε ότι το επόμενο διάστημα θα αναμένουμε θετική πρόοδο προς την κατεύθυνση της πιο στενής συνεργασίας με τις τρίτες χώρες. Ε, πραγματικά σας ευχαριστώ και ε, εύχομαι και η επόμενη Προεδρία, η Ιρλανδική Προεδρία, πάλι από μια χώρα που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, να μπορέσει να σταθεί αντάξια και να συνεχίσει τα καλά αποτελέσματα που εσείς φέρατε αυτή την περίοδο. Ευχαριστώ πολύ. Mr. Στον κυριο Παπαρικολάου, κύριο Το Πρόεδρε, ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους δύο Υπουργούς της Κυπριακής Δημοκρατίας για τον απολογισμό της εργασίας που έχουν κάνει κατά τη διάρκεια της ε, Κυπριακής Προεδρίας. Πράγματι έχει επιτευχθεί αρκετή πρόοδος σε πολλούς τομείς. Έχουν εξευρεθεί κοινέ συνισταμένες, παρόλο που εμείς ως ομάδα της αριστεράς διαφωνούμε αρκετά με την τελική θέση και του Κοινοβουλίου και έχουμε ε, καταψηφίσει ορισμένα πράγματα, αλλά αυτό δεν μειώνει καθόλου την ε, σκληρή δουλειά που έχει γίνει από τους ε, δύο Υπουργούς. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα της αλληλεγγύης και θα ήθελα να σταθώ λίγο στα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία θεωρώ απαραίτητα για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων. Είχαμε πρόσφατα ως ΛΥΠΕ επισκεφθεί την Ελλάδα, για παράδειγμα, και έχουμε δει πόση σημαντική πρόοδος έχει γίνει ακριβώς επειδή υπήρχαν αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και θα παρακαλούσα ιδιαίτερα την κυρία Μαύρου που έχει αναφερθεί ε, στα διάφορα ταμεία όπως το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης ε, να βεβαιωθεί ότι θα υπάρξει αρκετή, ε, αρκετό κονδύλι για να μπορέσουν αυτά τα, ε, τα ταμεία να συνεχίσουν να βοηθούν. Ξέρω ότι οι καταστάσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες, οι οικονομικές, αλλά αναμένουν πάρα πολλές ε, χώρες να βοηθηθούν οικονομικά για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που υπάρχουν σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τα κέντρα υποδοχής, τις διάφορες διαδικασίες κλπ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θέλετε να λάβετε το λόγο. Δύο ακόμα μιλητές. Ο κύριος έχει το λόγο πρώτος. <clears throat> Σας ευχαριστώ. Είχα ήδη ζητήσει το λόγο. Ίσως δεν με είδατε, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Κυπριακή Προεδρία για το έργο της εξορώματος της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπήρξαν παρουσιάσεις και προηγουμένων προεδριών που έχουμε παρακολουθήσει και έχουμε διαπιστώσει ότι μέσα σε ένα εξάμεινο είναι δυνατόν να αναλάβει μια προεδρία ευθύνη για πάρα πολλά θέματα, για τα θέματα εσωτερικών και δικαστικών ζητημάτων. Είδαμε να υπάρχουν βέβαια και σημεία εμπλοκή στον τομέα αυτοεργασίας. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορείτε να διεκπαιρεώσετε το πρόγραμμά σας και το γνωρίζουμε αυτό από το παρελθόν είναι μέσα από προσπάθειες υπέρβασης αυτών των εμπλοκών. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ και φυσικά υπάρχουν και κάποιες προτεραιότητες κομβικές για την πολιτική μας ομάδα, τις οποίες συμμεριζόμαστε και με άλλες πολιτικές ομάδες. Η κυρία Κάρμεν Ρομέρο, η συνάδελφός μου, νομίζω εντόπισε κάποιες από αυτές τις δύο σαφείς προτεραιότητες για την ομάδα των σοσιαλιστών και δημοκρατών. Μία από αυτές, με κίνδυνο να είμαι επαναληπτικός, μία από αυτές είναι η οδηγία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, η οποία θα παρουσιαστεί στις 10 Ιανουαρίου στην Επιτροπή μας και αναφερόμενος ιδίως στον κύριο Λουκά. Εδώ η κύρια μέρημνά μας προέρχεται από το γεγονός ότι στο Συμβούλιο έχουμε δει πολλές ανησυχίες, όχι απλώς μια στάση εμπλοκής, αλλά και πολλές ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο Έχουμε ανησυχίε εμεί μάλλον για τον τρόπο που αντιμετωπίζει το Συμβούλιο αυτή την οδηγία. Υπάρχει μια εξαίρεση του δημοσίου τομέα και μια σημαντική αλλαγή του πνεύματος του κανονισμού αυτού και της οδηγίας. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω από τον κύριο Λουκά ποια είναι η δική του άποψη για την μεταλαμπάδευση, για την μεταφορά μάλλον της κοιτάλης στην Ιρλανδική και Προεδρία για το θέμα αυτό που πιστεύω ότι και αυτή θα το αντιμετωπίζει σαν μια κύρια προτεραιότητα. Και όπως επίσης είπε η Κάρμεν προηγουμένως, υπάρχει οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου και ο τρόπος που έχει αντιμετωπιστεί από το Συμβούλιο και με την ε, με το νομοθέτημα για τη Eurodac που πέρασε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χθε, πάλι έχουμε κάποιε ανησυχίε για τη θέση του Συμβουλίου σε σχέση με όλα αυτά. Είναι φανερό ότι εσεί θα εγκαταλείψετε την Προεδρία, αλλά θα με ενδιαφέραν οι γενικέ σα απόψει για το πώ θα προχωρήσουν αυτά τα θέματα και με την Ελλαδική Προεδρία. Τέλο, αντιμετωπίσετε για τα τελικά τμήματα του πακέτου μετανάστευση μετά από τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν είναι προτεραιότητα της Προεδρίας ή ουσιαστικά δεν είναι προτεραιότητα κανενός για τους εργαζόμενους που περνά από μια επιχείρηση σε μια άλλη και για τους εποχιακούς εργαζόμενους. Αλλά το θέμα της ε, ε, μη τακτικού χαρακτήρα μετανάστευσης είναι ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Θα θέλαμε να ξέρουμε ποιες είναι οι προοπτικές για να υπάρξει περαιτέρω στα θέματα αυτά. Πιστεύω ότι οι προσπάθειες της Κυπριακής Προεδρίας μπορούν να είναι πρόσφορες για να προχωρήσει το θέμα αυτό, αλλά θα ήθελα να ακούσω και τις δικές σας απόψεις σχετικά. Ευχαριστώ κύριε Μωράης. Κυρία Παπαδοπούλου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχα ζητήσει και εγώ τον λόγο ε, και εγώ με τη σειρά μου να πω ότι ε, έχω δει την Κυπριακή Προεδρία αυτό το εξάμεινο να εργάζεται σκληρά για να ελοπίσει του στόχου τη και ο βασικό στόχο ήταν για μια καλύτερη Ευρώπη. Από την αναφορά που έχει γίνει από του δύο υπουργού και την κυρία Μαύρου και τον κύριο Λουκά, εκείνο το οποίο προσωπικά βλέπω είναι ότι δόθηκε έφαση σε θέματα τα οποία αφορούν ε, κοινωνική πολιτική, θέματα εμπορία προσώπων και χαίρομαι γιατί το Συμβούλιο νιοθέτησε συμπεράσματα και οργανώθηκε συνέδριο. Έκλεισε ο φάκελο για το citizenship, του Ευρωπαϊκού Έτο Πολιτών. Ε, Ω εισηγήτρια, πρέπει να πω ότι είχα την εμπειρία να ξεκινήσει ο πρώτο τρίλογο με την Δανέζικη Προεδρία και να ολοκληρωθεί επί Κυπριακή Προεδρία. Και θεωρώ ότι είναι ένα φάκελο ο οποίο θα μα δώσει την ευχαίρεια το 2013 να αναδείξουμε τι είναι τα ωφελήματα τα οποία προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια Εκείνο που με ανησυχεί όμω ιδιαίτερα ότι είναι για το φάκελο αυτό έχει δοθεί μόνο ένα budget, ένα εκατομμύριο. Και αυτό είναι πάρα πολύ μικρό συγκριτικά με προηγούμενα άλλα ευρωπαϊκά έτη και δεν ρωτούμε ποια είναι η αντίληψη του Συμβουλίου και πώ μπορούν να δουλέψουν ώστε με τόσο μικρό budget να υπάρχουν πραγματικά ε, τέτοιε δράσει που να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτε για τα δικαιώματα του που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Χαίρομαι επίσης γιατί έγινε ένα πολύ καλό συνέδριο στην Κύπρο, το οποίο παρακολούθησα όσον αφορά τη βία στην οικογένεια και υπάρχει πρακτικά ένα αποτέλεσμα, ένα ευρωπαϊκό εχειρίδιο για καταπολέμηση της βίας. Και όπως ξέρουμε, επειδή είμαι και μέλο στην Επιτροπή ΦΑΜ, το θέμα της βίας εναντίον των γυναικών είναι πάρα πολύ πλατή και χρειάζονται συνολικέ δράσει. Το εγχειρίδιο θα βοηθήσει. Επίση, χαίρομαι γιατί για τα ναρκωτικά έχει γίνει μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για το 2013-2020 γιατί όντω χρειάζονται πολλέ ε, δράσει και συνέργεια. Το δικό μου ερώτημα επικεντρώνεται και είναι ένα γενικό ερώτημα. Έχω δει ότι σε αρκετού φακέλου η Κύπρος προσπάθησε πολύ, γιατί είναι ένα μικρό παίχτη στην πολιτική σκακέρα και υπήρξε όντω ένα έντιμο διαμεσολαβητή. Πολλοί φάκελοι έφτασαν σχεδόν στο παραπέντε για να κλείσουν. Ποια ήταν τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν. Ήταν γιατί υπάρχουν διαφορετικές απόψεις από μεγάλες χώρες μέσα στο Συμβούλιο, οι οποίες είχαν δικά τους εθνικά συμφέροντα να εξυπηρετήσουν. Θέλω να είστε λίγο πιο ξεκάθαροι. Ποια ήταν τα πραγματικά εμπόδια που βρέθηκαν εντός Συμβουλίου για να μην κλείσουν φάκελοι που ήταν κοντά στο να κλείσουν. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. No more hands. Δεν βλέπω κανένα άλλο ομιλητή. <coughs> Ερχόμαστε τώρα στις απαντήσεις και από τους δύο υπουργούς. Μπορούμε να αναστρέψουμε τη σειρά ή θέλετε να ακολουθήσουμε την ίδια σειρά. Κύριε Μαύρου, έχετε το λόγο πρώτη. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, παρατηρήσεις, για τις ερωτήσεις και για τα καλά σας ε, λόγια. Ε, σε ό,τι αφορά τις ε, παρατηρήσεις της ε, κυρίας Ρομέρο Λόπες για το ε, κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, ε, ναι, το σύστημα του Δουβλίνου είναι περίπλοκο. Ναι, το, στο Eurodac υπάρχουν επιφυλάξεις και από κράτη-μέλη και από μέλη του, Ευρωκοινο... Ευρωκοινοβουλίου και από όλες τις συνιστώσεις. Όταν ξεκινούσε πριν από χρόνια αυτή η προσπάθεια για το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, κανείς δεν πίστευε ότι θα ήταν εύκολος ο δρόμος. Ε, έπρεπε να βρεθούν ε, οι, ε, οι συμβιβασμοί και οι κοινέ συνισταμένες ε, μεταξύ πολλών διαφορετικών συνιστώσεων. Ε, εκείνο που θα έλεγα ότι ε, έχουμε διαφορετική εκτίμηση ε, είναι η άποψη ότι δεν πήγαμε ένα βήμα μπροστά. Αντίθετα, θα έλεγα ε, όχι μόνο το γεγονός ότι έχει υπάρξει ήδη συμφωνία για τον κανονισμό του Δουβλίνου, για την οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής, για το γεγονός ότι στην οδηγία ε, για τις ε, διαδικασίες έχουμε φτάσει ε, νομίζω στο τέλος με λίγη ακόμα προσπάθεια μπορεί να βρεθεί συνδυασμός Για το Eurodac επίσης μπορούμε να βρούμε τις ισορροπίες μεταξύ της προστασίας των ατόμων και της εξυπηρέτησης των εθνικών συμφερόντων και της καταπολέμησης των καταχρήσεων του συστήματος ασύλου. Εάν δούμε το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου με τη μορφή που έχει πάρει τώρα μετά από τις ε, διαπραγματεύσεις όλες, νομίζω όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι από τη μια παρέχει ένα ψηλότερο επίπεδο προστασίας σε εκείνους που πραγματικά το έχουν ανάγκη από τη υφιστάμενη κατάσταση γιατί με αυτό είναι που πρέπει να συγκρίνουμε, όχι με, με το πώς θα θέλαμε να είναι το σύστημα, ο κάθε ένας από εμά ξεχωριστά. Άρα παρέχει από τη μια ένα ψηλότερο επίπεδο προστασίας, ε, ένα πιο, μια πιο συγκροτημένη διαδικασία ε, για την εξέταση των αιτήσεων και την παροχή ασύλου και μια ομοιόμορφη αντιμετώπιση των αιτητών προστασίας σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουμε ότι το γεγονός ότι δεν υπήρχε ομοιομορφία ε, ήταν ταυτόχρονα και παράγοντας που ενεθάρρυνε τις καταχρήσεις ε, του συστήματος. Ε, έχουμε κάνει, θα έλεγα, πολλά βήματα μπροστά. Ε, ως ε, το ευρωπαϊκό τούτο ε, οικοδόμημα. Ο καθένας βέβαια διατηρεί τις απόψεις και τις επιθυμίες του. Αλλά νομίζω γνωρίζετε καλύτερα από πολλούς ότι καταλήγουμε στο τέλος σε συμφωνίες μέσα από μια σειρά συμβιβασμών ο καθένας του. Αναφέρθηκε η κυρία Παπαδοπούλου γιατί ενώ είμαστε στο παραπέντε ε, δεν ε, έχουμε ε, καταφέρει να καταλήξουμε σε συμφωνία. Πρώτα-πρώτα γιατί ήταν ένας πολύ φιλόδοξος στόχος και ένα περίπλοκο σύστημα. Χαρακτηριστικά απαντώντας στην ίδια ερώτηση η Επίτροπος Μάλμστρομ πριν δέκα μέρες είπε ότι αν με ρωτούσατε πριν ένα χρόνο, έξι μήνες, αν θα καταλήγαμε σε συμφωνία μέχρι το τέλος του 12, θα σας έλεγα αποκλείεται. Το γεγονός ότι αυτούς τους μήνες ε, δουλέψαμε πολύ σκληρά και με πολύ ειλικρίνεια, λαμβάνοντας υπόψη και συμφέροντα κρατών μελών, και ανησυχίες κρατών μελών, ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες ε, της οικονομικής ύφεσης. Αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τις αξίες τις οποίες ήθελε να υπερασπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από αυτό το κοινό σύστημα ασύλου, ε, νομίζω ότι ε, καταφέραμε να γεφυρώσουμε ένα μεγάλο χάσμα για να είμαστε σήμερα εδώ έστω στο παραπέντε ε, να καταλήξουμε. Ε, η, απαντώντας και στον κύριο Μωράες πού πάει το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, ε, πρέπει να σας πω ότι η μόνη μου έγνοια ε, είναι να μην αφήσουμε την δυναμική που έχει δημιουργηθεί να χαθεί. να μην αφήσουμε το, τις οικονομικές δυσκολίες ε, να μας εμποδίσουν από το να, ε, να βάλουμε στόχους για, μια, για ένα καλύτερο σύστημα ε, προστασίας. Ε, είμαι βέβαιη ότι η Ιρλανδική Προεδρία θα παραλάβει τη σκητάλη και θα δουλέψει με την ίδια επιμονή ε, και ελπίζω με την ε, βοήθεια όλων ε, πολύ σύντομα να μπορούμε να μιλούμε για ολοκλήρωση της προσπάθειας αυτής. Σε ό,τι αφορά την αναφορά της κυρίας Ρομέρο Λόπες για τις συμφωνίες, σας είπα ότι για μας ο διάλογος και η συνεργασία με χώρες γειτονικές, χώρες προέλευσης ε, μεταναστών ε, είναι ε, βασική πολιτική επιλογή. Σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες, για μεν την Ινδία έχει υπάρξει καταρχήν απόφαση για την κοινή ατζέντα για την κινητικότητα και τη μετανάστευση και θεωρείται πραγματικά επιτυχία αυτή η συμφωνία ε, λόγω της πρωτοπόρας φύσης του εχειρήματος, ε, του μεγέθους της χώρας, οι σχέσεις με την οποία είναι περίπλοκες σε αρκετά θέματα. Είναι η πρώτη ε, φορά στα ιστορικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λαμβάνεται απόφαση για εγκαθίδρυση αυτού του προγράμματος συνεργασίας με τρίτη χώρα που αποτελεί στρατηγικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα είναι καταρχήν ε, συμφωνία, ε, τα κείμενα τα επεξεργάζεται ακόμα η ομάδα. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα εργασίας ε, με τη Ρωσία για την επόμενη διετία, έχουμε καταλήξει, υπάρχει επίσημο έγγραφο, το οποίο είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου ε, ενώ για τις ε, συμφωνίες εταιρικής σχέσης κινητικότητας με το Μαρόκο και την, ε, Ισία οι διαπραγματεύσεις ουσιαστικά είναι στο τελικό τους στάδιο. υπολογίζουμε ότι η ομάδα εργασίας θα μπορεί να καταλήξει σε τελικό έγγραφο πολύ σύντομα. Κύριε Παπα-Νικολάου, αυτά εν ολίγης απαντούν ε, και στο δικό σας ε, ερώτημα, παρόλο που, όπως έχω πει, ε, έχουν γίνει τέτοιες προσπάθειες με πολλές άλλες χώρες. Γίνονται επαφές με την Ιορδανία, για παράδειγμα, με την Κίνα, ενώ έχουμε ε, προωθήσει και τον διάλογο Ευρωπαϊκής Ένωσης Λατινικής Αμερικής, Καραϊβικής, Ασίας ε, κλπ. Η Τουρκία έχει απασχολήσει ε, ιδιαίτερα το Συμβούλιο στα πλαίσια των, των συζητήσεων για την ιδιαίτερη σχέση της χώρας αυτής με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ε, συζητήσει την ε, προοπτική στο μέλλον εγκαθίδρυσης ενός ειδικού συστήματος μια ιδιαίτερη σχέση όσον αφορά τις θεωρήσεις. ταυτόχρονα όμως μας προβληματίζει το γεγονός ότι από την χώρα αυτή βλέπουμε ε, να, ε, να περνούν σημαντικά ε, παράνομα μεταναστευτικά κύματα και είμαστε σε επαφή μέσω ιδιαίτερα των προσπαθειών που καταβάλει η Επιτροπή για πιο αποτελεσματική διαχείριση των φαινομένων αυτών η συνεργασία με τις γειτονικές χώρες ευρύτερα θεωρώ ότι απαντά και σε αυτό το ε, πρόβλημα ε, που είναι σημαντικό. Ε, βεβαίως το, στην όλη προσπάθεια νομίζω συμβάλλει ε, και η προσπάθεια για ρύθμιση της νόμιμης μετανάστευσης. Κύριε Μωράες, ε, μπορεί ε, η σύμβαση για τους εποχικά εργαζόμενους ε, να μην θεωρείται από κάποιους προτεραιότητα. Σας διαβεβαιώνω ότι ως Προεδρία ε, δουλέψαμε με πολλή επιμονή και για τις δύο οδηγίες που καλύπτουν την νόμιμη μετανάστευση Χαίρομαι γιατί με τη δική σας την ε, βοήθεια καταφέραμε να ξεκινήσουμε με ένα καλό τρίλογο και αν και τα πράγματα φαίνονταν πολύ δύσκολα πριν ε, λίγους μήνες, ε, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε ένα καλό στάδιο και σας ευχαριστούμε. Έτσι κι αλλιώς τα θέματα μετανάστευσης είναι όπως ένα puzzle. Ε, κάθε προσπάθεια που κάνουμε βάζει ένα κομματάκι της εικόνας. Δεν υπάρχει τρόπος να, ε, να διαχειριστούμε ε, όλα τούτα τα ζητήματα με ένα ομοιόμορφο και απόλυτο τρόπο. και τέλος, στα θέματα των ταμείων, όπως έχουμε πει, κύριε Τρενταφυλλίδη, ε, ε, είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που έχουμε καταφέρει να... time, so we... Δεν έχουμε χρόνο, κύριε Υπουργέ. Θα πρέπει να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Λουκά για να απαντήσει. Επομένω, αν μπορείτε να συνοψίσετε. Σας ευχαριστώ και των προτέρων. Εντάξει. Θα αναφερθώ στο Ταμείο. Για το Ταμείο ε, Εσωτερικής Ασφάλειας Συνόρων και Θεωρήσεων και για τον Οριζόντιο Κανονισμό, νομίζω πολύ σημαντικά ε, είναι και η συμφωνία για τα προγράμματα SOLID, για τα κράτη που ε, έχουν δεχθεί βοήθεια από τον μηχανισμό στήριξης. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι ε, τα τελικά αποτελέσματα στον τομέα αυτό θα εξαρτηθούν από τα γενικότερα αποτελέσματα στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Minister. Now... Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Τώρα η σειρά σας κύριε Λουκά. Πολύ σύντομος κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ αν μπορείτε να αναφερθείτε επί τόσο συγκεκριμένο σημείο γιατί δεν έχουμε χρόνο. Θα ήθελα να, να απαντήσω στην κυρία Λόπες και να πω ότι ε, έχει δίκιο ότι έχω παραλείψει στην προσπάθεια μου να συντομεύσω την αρχική μου ομιλία, ενημέρωση ε, για το θέμα της οδηγίας. Ε, με βάση τη συνθήκη τη Λισαβόνα, οι κανόνε προστασία προσωπικών δεδομένων πρέπει να τη χάνουν ομοιόμορφη εφαρμογή σε όλου του πρώην πυλώνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτόν η Προεδρία θεώρησε σημαντικό να αφιερώσει κατά αναλογία περισσότερο χρόνο στη συζήτηση του γενικού κανονισμού, αφού οι βασικέ αρχέ αυτού θα πρέπει να κατανοηθούν και να συμφωνηθούν πριν ενσωματωθούν στην οδική, ειδική οδηγία. Τόσο για τον κανονισμό όσο και για την οδηγία υποβλήθηκαν από τα κράτη-μέλη γραπτά σχόλια επί των άρθρων που καλύφθηκαν. Για τον κανονισμό ετοιμάστηκε ένα δεύτερο προσχέδιο το οποίο θα παραδοθεί στην Ιρλανδική Προεδρία για περαιτέρω νομοτεχνική επεξεργασία. Τα πιο πάνω καταγράφηκα στην έκθεση προόδου που η Κυπριακή Προεδρία υπέβαλε στο Συμβούλιο Δικαιοσύνη και Εσωτερικών Υποθέσεων τον Δεκέμβριο. Ειδικά για το, για το ερώτημα σας για την πρόταση οδηγία σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως έχω αναφέρει προηγουμένως, στο Συμβούλιο ΔΕΗ του Δεκεμβρίου εγκρίναμε την έκθεση πρόοδου. Όπω έχουμε δηλώσει επανειλημμένα για την Κυπριακή Προεδρία, το θέμα να αποτέλεσε προτεραιότητα και αντιμετωπίστηκε ω ένα πακέτο. Ακριβώ για αυτόν τον λόγο παρουσιάσαμε ενώπιον των Υπουργών μια ενιαία έκθεση πρόοδου η οποία καλύπτει και τα δύο νομοθετήματα. Ω προ το Πώ βλέπουν τα κράτη-μέλη την πρόταση για την οδηγία, δεν μπορούμε να πούμε πολλά γιατί δεν έγιναν διευρυμένε συζητήσει. Δεν θα αρνηθώ ότι ένα αριθμό κρατών μελών ήγηραν ορισμένα προβλήματα όσον αφορά ορισμένε ουσιαστικέ επιλογέ πολιτική εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν τέθηκε ποτέ σε επίπεδο του Συμβουλίου θέμα απόσυρση ή τερματισμού των εργασιών για την οδηγία. Όπω έχετε ακούσει, δεν έχω ξεχάσει την οδηγία. Έχουμε ήδη αφιερώσει αρκετό χρόνο σε τεχνοκρατικό επίπεδο και προγραμματίζουμε περαιτέρω συζήτηση του θέματο αποκλειστικά επί τη πρόταση οδηγία αύριο και πεθαύριο» στην αρμόδια οργασία, ομάδα εργασία DAPIX. Ξεκίνησε ε, κατάρθρο συζήτηση και έχει καλύψει τα άρθρα 4 ως 8. Ελπίζουμε ότι αυτή, σε αυτήν τη διήμερη συνάντηση, καθώ και το γεγονό ότι τα κράτη-μέλη έχουν ανταποκριθεί στο αίτημα τη Προεδρία για να στείλουν τα σχόλια του επί τη οδηγία, θα προωθήσουμε περαιτέρω την εργασία που γίνεται. Κάποια από τα σχόλια που έχουμε λάβει αναφέρονται στο έργο που, έχουν ήδη, που έχει ήδη επιτελεστεί από την πρόταση κανονισμού. Συνεπώ, η εργασία που έχει γίνει επί του κανονισμού ουσιαστικά διευκολύνει και θα επιταχύνει τι συζητήσει επί τη οδηγία. Όσον αφορά το θέμα της προσχώρησης της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως έχω ήδη προηγουμένως αναφέρει. Οι διαπραγματεύσεις έχουν επαναρχίσει και, ε, και έχουν λάβει χώρα τρεις γύρι διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αναφορικά με το πακέτο για τα δικονομικά δικαιώματα και ιδιαίτερα όσον αφορά το θέμα νομικής αρρωγής, αναμένεται η κατάθεση της σχετικής οδηγίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, η κυρία Λοπές αναφέρθηκε ε, στην επιχείρηση Αφροδίτη. Τα αποτελέσματα της επιχείρησης αυτής παρουσιάστηκαν στην ομάδα εργασίας για την ε, αστυνομική συνεργασία και μπορώ να πω ότι η συμμετοχή και η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών ήταν εξαιρετική. Λεπτομέρειες για την επιχείρηση αυτή μπορούν να σας σταλούν στο γραφείο σας πολύ σύντομα. Ε, θα ήθελα και πάλι κύριε Πρόεδρε να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ειδικά την Επιτροπή ΛΥΠΕ και τους εισηγητές για την άψογη συνεργασία που είχαμε σε θέματα ε, εσωτερικών και δικαιοσύνης. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και τους δύο, κυρία Μαύρου και κυρία Λουκά, για τις προσπαθίες σας και για την ε, δέσμευσή σας ε, έτσι ώστε να γεμίσετε με επιτυχία στο εξάμεινο της ε, Κυπριακής Προεδρίας. Σας ευχαριστούμε που περιβρεθήκατε εδώ για να μας παρουσιάσετε όλα αυτά τα ζητήματα και για την προσπάθεια που κάνετε να συνοψίσετε και να απαντήσετε στα σχόλια των μελών της Επιτροπής Λίβης. Σας ευχαριστούμε λοιπόν, Περιβρεθήκατε εδώ, θα συνεχίσουμε με τη μέση διάταξη.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 So, now. Να περάσουμε στο σημείο 17, την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 7η έκθεση, σχετικά με τη διατήρηση από ορισμένες τρίτες χώρες υποχρεώσεων θεώρησης κατά παράβαση της αρχής της αμοιβαιότητας. Θα καλωσορίσουμε τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μας παρουσιάσουν την 7η έκθεση. και θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Ντεκόιστερ για να μας παρουσιάσει αυτό το σημείο. Thank you, Mr. Ευχαριστώ. Είναι ικανοποίησή μου να βρίσκομαι εδώ σήμερα για να σας παρουσιάσω την 7η έκθεση αμοιβαιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υιοθετήθηκε στα τέλη Νοεμβρίου η αμοιβαιότητα είναι ένα δύσκολο θέμα. Βρίσκεται δύο φορές στην ημερησία διάταξη της Επιτροπής σας. Καταρχήν έχουμε την 7η έκθεση της ε, και κατόπιν θα συζητηθεί ως ε, τμήμα τη τροπής του κανονισμού που τροποποιεί τον κατάλογο των ε, θεωρήσεων. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητήθηκε διεξοδικά και μπορεί να καταλήξουμε σύντομα σε συμφωνία. Η 7η έκθεση εμβιότητας έπρεπε καταρχήν ε, να παρουσιαστεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου φέτος, ε, μέχρι τις 30 Ιουνίου, αλλά η Κομπισιόν ε, ανέβαλε τη διαδικασία για δύο μήνες περίπου, προκειμένου μέχρι τα τέλη του έτους να παρουσιάσει μια σαφή εικόνα της κατάστασης, της μη αμοιβαιότητας που αφορά τις τρίτες χώρες ελπίζουμε αυτή τη στιγμή ότι ο νέος μηχανισμός ε, αμοιβαιότητας να υιοθετηθεί. Πιστεύω ότι όλα τα όργανα συμφωνούν ότι ο μηχανισμός αμοιβαιότητας ε, θα πρέπει να καταστεί πιο αποτελεσματικός. Και αυτό είναι και θέμα στην απογευματινή μας ε, συζήτηση. Αυτό τώρα σημαίνει δεν έχει λειτουργήσει καλά το σημερινό σύστημα, δεν ήταν αποτελεσματικό. Όλα αυτά εξαρτώνται από ποια σκοπιά θα το δείτε. Υπήρξε μια περίπτωση όπου μια χώρα επανεσύγα για την απέτηση θεώρησης ε, για πολίτες ενός κρατούς μέλους. Έχουμε την υπόθεση Καναδά-Τσεχίας. Η περίπτωση αυτή της μη αμοιβαιότητα εξακολουθεί να υπάρχει. Αν δείτε λοιπόν την επιτυχία του μηχανισμού αμοιβαιότητα, λαμβανοντα υπόψη την εισαγωγή απέτησης ε, ε, θεωρήσεων θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για αποτυχία. Αν δείτε όμως ε, τις υποθέσεις που υπήρχαν τη στιγμή που κατέστη εφαρμοστέο το σημερινό σύστημα, το νέο σύστημα, μπορούμε να πούμε σήμερα ότι είναι αποτελεσματικό επειδή έχει επιλύσει αρκετές υποθέσεις. Όταν ε, άρχισε να εφαρμόζεται ο μηχανισμο 2005 2005-2006, είχαμε περίπου 100 υποθέσεις μη αμοιβαιότητες με 18 χώρες. Ε, σήμερα παραμένουν πολύ λίγες περιπτώσεις με δύο σημαντικούς εταίρους, τι ΗΠΑ και τον Καναδά. Σήμερα το απόγευμα λοιπόν θα συζητήσουμε πώς μπορεί να καταστεί πιο αποτελεσματικός ο μηχανισμός, όμως τώρα θα σας δώσω θα σας κάνω μια σύντομη επισκόπηση του τι συνέβη της πρόοδου που έχει σημειωθεί από την τελευταία έκθεση της Κομισιόν το Νοέμβριο του 2010. Η πρώτη επιτυχία που μπορούμε να αναφέρουμε έχει να κάνει με τη σχέση με τη Βραζιλία. Εδώ, φέτος τον Οκτώβριο, τέθηκε σε ισχύ η αμοιβαία συμφωνία άρσης υποχρεωση θεωρησίων για τους κατόχους κανονικών διαβατηρίων. Έτσι λοιπόν έληξε μια κατάσταση μια αμοιβαιότητας για πολίτες της Κύπρου, της Εστονίας, της Λετωνίας και της Μάλτας για τέσσερα κράτη-μέλη. Έτσι λοιπόν έχει επιληθεί αυτό το ζήτημα, έχει λήξει. Κατόπιν έχουμε την κατάσταση με την Ιαπωνία, όπου η Ρουμανία μέχρι πριν 2-3 χρόνια ήταν υπό υποχρεώση θεώρησης, ε, χάρη σε όλες τις δράσεις που αναλήφθηκαν, η Ρουμανία απέκτησε μια προσωρινή άρση θεώρησης από την Ιαπωνία και τώρα είμαστε σε επαφή και με τις δύο αρχές, ρουμανικές και ιαπωνικές, για να αποκτήσουμε μία ε, απόφαση από την κυβέρνηση της Ιαπωνίας, είτε να παρατείνει αυτή την προσωρινή άρση υποχρεωσιτόρησης για τους πολίτες της Ρουμανίας ή να τους ε, προσφέρει μια οριστική απαλλαγή. Κάτι άλλο, ίσως λιγότερο θεματικό, μια άλλη σημείωση πρόοδου ήταν με τον Μπρουνέη οι πολίτες των κρατών μελών ε, ήδη εποφελούνταν ε, από απαλλαγή θεώρησης για παραμονές μέχρι 90 ημέρες. Όμως οι πολίτες ε, των συνδεόμενων χωρών Σέγγεν επίσης είχαν απαλλαγή υποχρέωσης θεώρησης, αλλά μόνο για διαμονή μέχρι 30 ημέρες ή μόνο για 14 ημέρες. Τώρα το Μπρουνέ επιβεβαίωσε ότι η απαλλαγή υποχρέωσης θεώρησης για αυτές τις συνδεόμενες χώρες έχει ε, παραταθεί μέχρι τις 90 ημέρες. Έτσι λοιπόν το μόνο που παραμένει να γίνει εδώ είναι να διασφαλίσουμε ότι και το Λιχτενστάιν και οι πολίτες του υποφελούνται από μια τέτοια απαλλαγή για παραμονές μέχρι 90 ημέρες Δεν ξέρω βέβαια πόσοι από το Λιχτενστάιν θα ταξιδέψουν τώρα στο Πρινέ για να παραμείνουν από ένα ως τρεις μήνες, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να συνεχίσουμε αυτές τις προσπάθειες. Είναι βέβαια πολύ μικρή περίπτωση μια αμοιβαιότητας ε, που αφορά ε, τις ημέρες, τη διάρκεια της παραμονής. Και κατόπιν έχουμε τα δύο κυρία ζητήματα που εξακολουθούν να είναι επιτάπητος με τον Καναδά και τις Ηνωμένε Πολιτείε. Εδώ για τις Ηνωμένε Πολιτείε εξακολουθούν να υπάρχουν ε, τέσσερι χώρες για τις οποίες απαιτείται για τους πολίτες των οποίων απαιτείται θεώρηση και για τον Καναδά τρία κράτη-μέλη. Και φυσικά η Κομισιόν έχει έρθει σε επαφή με τις αρχές των ΗΠΑ και συνεχίζουμε να τονίζουμε ότι χρειαζόμαστε πλήρη αμοιβαιότητα, δηλαδή ότι πρέπει να αποκτήσουμε απαλλαγή υποχρέωση θεώρηση και για τους πολίτες της Κύπρου, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας. Τώρα, να σας αναφέρω κάποια στοιχεία για την κατάσταση με τις ΗΠΑ. Ξέρετε ότι υπάρχει απέτηση θεώρησης και υπάρχει ένα σύστημα ΕΣΤΑ για όσους ε, απαλλάσσονται από υποχρεώσεις θεώρησης θα πρέπει να ζητήσουν μια ηλεκτρονική άδεια ταξιδίου. Η Κομισιόν ε, αξιολογεί σε μια έκθεση για το αν αυτή η ΕΣΤΑ είναι μια μεταμφιεσμένη θεώρηση. Αν δηλαδή αυτή η διαδικασία ισοδυναμεί με θεώρηση και κατόπιν ε, θα ξέρει κάποια συμπεράσματα. Η Κομισιόν ε, βέβαια πάντα δήλωνε ότι την ε, έκθεση αυτή ε, θα την καταρτήσει όταν έχουμε τον οριστικό κανόνα για την ΕΣΤΑ και αυτός ο κανόνας δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί από τις Αμερικανικές Αρχές. Αυτό είναι κρεμέ ζήτημα λοιπόν ακόμη. Τώρα, τι θα μπορούσε να μας δώσει κάποια ελπίδα για να επιλύσουμε για αυτά τα τέσσερα κράτη-μέλη ε, τα προβλήματα είναι ότι υπάρχουν ε, πολλά νομοσχέδια στο Κογκρέσο, τον είπα, με στόχο να διευκολύνουν τις συνθήκες πρόσβασης ε, στο πρόγραμμα απαλλαγής υποχρεώσεις θεώρησης. Επίσης είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ο πρόεδρος Ομπάμα υποστήριξε αυτά τα νομοσχέδια και Νομίζω ότι ήταν αυτό πλέον έκτιμα για το πρόγραμμα απαλλαγή υποχρέωση θεωρήση ότι είχαμε την επανεκλογή του κ. Μπαμά. Φυσικά υπάρχουν και άλλα πλέον γενικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ε, γενικά δείχνει κατανόηση ε, και είναι υπέρ του να επεκταθεί το πρόγραμμα και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Και μια άλλη θετική εξέλιξη είναι η τάση στι ΗΠΑ να αρχίσουν ε, να προωθούν τον τουρισμό μέσω διευκόλυνσης θεωρήσεων και μέσω νέων απαλλαγών ρώσης θεώρησης για να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη. Ένα άλλο υποδόμα είναι η λεγόμενη προσέγγιση του track, η δίτη προσέγγιση. Ξέρετε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, στην νομοθεσία τη θέτει μία σειρά προποθέσεων για την πρόσβαση στο πρόγραμμα απαλλαγή θεώρηση. Παραδείγματο χάρη, η ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα θα πρέπει να εκδώσει βιομετρικά διαβατήρια. Ξέρετε ότι έχουμε ένα κανονισμό που επιβάλλει στα κράτη-μέλη να εκδώσουν βιομετρικά διαβατήρια. Έτσι λοιπόν μέσω της εφαρμογής του κανονισμού αυτού οι σχετικέ προποθέσει πληρούνται για την απαλλαγή τη υποχρέωση θεώρηση. Έτσι λοιπόν είχαμε κάποια στιγμή αυτή την ε, ε, διπλή παράλληλη προσέγγιση όπου υπήρχε ένα μνημόνιο κατανόηση ε, με τι ΗΠΑ ότι οι συνθήκε απαλλαγή υποχρέωση θεώρηση που θα ήταν στο πρώτο πυλώνα, δηλαδή βιομετρικά, διαβατήρια και ασφάλεια τη αεροπλία, θα θεωρούνται από τις ΗΠΑ ότι πληρούνταν αν εφαρμόζονταν η νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερο επίπεδο, δηλαδή τρίτος πυλώνας, έχουμε την τρομοκρατική συνεργασία και ε, τη συνεργασία μεταξύ ιδιωτικών αρχών. Διμέρει σχέσεις λοιπόν των κρατών μελών με τις Ηνωμένες Πολιτείες ως μια άλλη προϋπόθεση που πρέπει να πληρείται ε, προκειμένου να συμμετέχουν οι χώρες, να μπορούν να μπουν ή να παραμείνουν στο πρόγραμμα απαλλαγής και κατόπιν αιτήματο ε, του Κοινοβουλίου αξιολογήσαμε αυτό το πρόγραμμα υπό το φως συνθήκης της Λισαβόνας και προσθέσαμε στην έκθεση συγκεκριμένο παράρτημα το οποίο λεπτομερώς εξηγεί και αναλύει τα αποτελέσματα και πιστεύουμε ότι αυτή η διπλή προσέγγιση αφού τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας εξακολουθεί να ισχύει Όμω, επίση ελέγξαμε αν οι διμερεί συμφωνίε που έχουν συναυθεί από τα κράτη-μέλη με τι Ηνωμένες Πολιτείες εάν το ευρωπαϊκό δίκαιο. Δηλαδή τα υφιστάμενα μέσα τρίτου πυλώνα για την ανταλλαγή πληροφοριών και την καταπλήρωση τρομοκρατίας και για τη συνεργασία των διοικητικών αρχών, την επιβολή του νόμου. Ήδη η Κομισιόν στην έκθεσή της δηλώνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων. Αν δείτε τη σημερινή απόφαση πλαισίου για την προστασία των δεδομένων από τη μορφή του τρίτου πυλώνα. Σας καλώ όλους προσεκτικά να διαβάσετε την έκθεση της Κομισιόν για το σημείο αυτό, γιατί έχει διατυπωθεί πολύ προσεκτικά. Δεν λέμε ότι τα κράτη-μέλη με τις διμερείς συμφωνίες ή ορισμένα από τα κράτη-μέλη παραβιάζουν ε, το ευρωπαϊκό δίκαιο για το θέμα αυτό. Υπάρχουν όμως ανησυχίες γιατί οι συμφωνίες δεν είναι πάντοτε σαφείς επί όλων των σημείων, όπως να το σχάρι ο περιορισμός του σκοπού, αλλά μπορώ να σας πω ότι μία πιθανή ε, αποκατάσταση αυτών των ε, ανησυχιών ε, ήδη συζητείται, όπως παίρνει το χάρη η διαπραγμάτευση της Συμφωνίας Ομπρέλας, που θα συμπληρώσει αυτές τις διμερείς συμφωνίες και θα διασφαλίσει ότι υπάρχουν όλες οι ασφαλιστικές δικλείδες που απαιτούνται. Τελευταίο σημείο για τις Ηνωμένε Πολιτείε. Στη νομοθεσία τους έχουν ορισμένες προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν ε, με ποσοστά περαιτέρω παραμονής και ποσοστό άρνησης χορήγησης θεώρησης. Και μπορώ να σας πω ότι αυτό το τελευταίο είναι 3% και μόνο η Κύπρος θα έφτανε σε αυτό το όριο. Οι άλλες τρεις χώρες είναι πάνω από αυτό το κατόφλι. Υπάρχουν ε, δυνατότητες ε, για το Υπουργείο εσωτερικό να αυξήσει αυτό το ποσοστό άρνησης θεωρησιών στο 10% αν ε, το σύστημα εξόδου αεροδρομίου θα λειτουργήσει, κάτι που θα μπορέσει να βοηθήσει το σύστημα να λειτουργήσει καλύτερα, Όμω, ε, τώρα συζητούμε πότε θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, το συζητούμε με τους Αμερικανού συναδέλφους, γιατί αν δείτε μόνο αυτά τα νούμερα, τότε θα επέτρεπε και στην Πολωνία να μπορέσει να μπει στο πρόγραμμα απαλλαγή θεώρηση. ενώ τα άλλα δύο κράτη θα έφταναν με το ποσοστό της περίπου σε αυτό το 10%. Και κάτι τελευταίο για τον Καναδά. Το θέμα Καναδά Τσεχική Δημοκρατίας είναι αυτό που νομίζω πέρσι οδήγησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο να προβεί σε δηλώσεις ότι πρέπει να καταστήσουμε πράγματι πιο αποτελεσματικό το μηχανισμό αβεβαιότητα. Τα όσα συνέβησαν τα δύο τελευταία χρόνια θα τα δείτε στην έκθεση. Έχουμε λεπτομερή επισκόπηση των συναντήσεων που έλαβαν χώρα. Α είμαστε σαφεί. Κάποια στιγμή, πριν δύο χρόνια, είχαμε συμφωνήσει σε μια σειρά μέτρων που θα επέτρεπε στον Καναδά να άρει την απέτηση θεώρησης ε, πριν, τεθείς πριν έχει τεθεί σε ισχύ. Ε, είναι νομοθεσία για το άσυλο, όμως τελικά δεν ε, ίσχυσε κάτι τέτοιο. Υπήρξε αύξηση ε, των ετούντων άσυλο στον Καναδά ε, με ψεύτικα κίνητρα ζήτουσαν άσυλο για να υποφεληθούν από ένα γενναιόδωρο σύστημα, παραδείγματο χάρη σε σχέση με τα επιδόματα που καταβάλλονται στου ετούντε άσυλο. Να σας ενημερώσω ότι πριν δύο-τρεις μέρες, στις 15 του μηνός, μία δεύτερη νομοθεσία περί ασύλου τέθηκε σε ισχύ στον Καναδά που θα μειώσει παραδείγματο χάρη δραστικά τη διάρκεια της διαδικασίας αίτησης ασύλου για τους αιτούντες άσυλο που έρχονται από ορισμένε χώρες που θεωρούνται ασφαλείς. Καθορισμένες χώρες, designated countries από τις ε, καναδικές αρχές θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ταχεία διαδικασία που θα διαρκούσε 30 με 45 μέρε ενώ σήμερα η διαδικασία, σύμφωνα με ενημέρωση από τις Καναδικές Αρχές, διαρκεί 600 ημέρε. Έτσι λοιπόν αυτό θα λειτουργούσε ω αποτρεπτικό και γι' αυτό η Κομισιόν πάντοτε δήλωνε ότι όταν αυτή η νομοθεσία τεθεί σε ισχύ, ο Καναδάς θα πρέπει να ρει την υποχρέωση θεώρησης καταρχήν για τους Τσέχους πολίτες και για τη Ρουμανία και για τη Βουλγαρία, αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Εξετάζουμε λοιπόν το ζήτημα, περιμένουμε να δούμε την εφαρμογή της νομοθεσίας για να ελέγξουμε ποια είναι τα αποτελέσματα, ποιο είναι ο αντίκτυπος επί του αριθμού των ετησίων ασύλου. σε αυτού. Ο Καναδάς επίσης ζητά συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη στο ζήτημα αυτό. Όπως στην περίπτωση Τσεχίας Καναδά και έχουμε και άλλους με το τεσάσιλο και πάλι έχουμε εδώ ένα παιχνίδι παραγόντων έλκυσης και όθησης. Τώρα, οι παραγόντες έλκυσης θα πρέπει να διευθετηθούν μέσω της νομοθεσίας για το άσυλο. Όμως ε, και κάποια μορφή τεχνικής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υπάρχει όταν επιστρέφονται κάποιοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενημερώνονται σωστά οι πολίτες για τις αλλαγές στην κρατική νομοθεσία περί ασύλου. Όμως η Κομισιόν, και τελειώνω πρόεδρε, πάντοτε τονίζει ότι τέτοιες μορφές συνεργασίας δεν θα πρέπει να γίνουν νέες προϋποθέσεις για να αρθεί η απέτηση υποχρεώσεις θεώρησης από τον Καναδά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κόιστερ. Έχουμε τώρα κάποια σημεία τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε πριν από τη συνάντηση των συντονιστών στο τέλος της ημέρας. Ε, Ε, αρχίζουμε τώρα τη συζήτηση και δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Άλβαρο πρώτα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση για τον μηχανισμό αμοιβαιότητος για τις προξενικές θεωρήσεις είναι ευρύτερη από την, ε, η συζήτηση αυτή από απλώς την άρση του μηχανισμού για τις προξενικές θεωρήσεις. Το Κοινοβούλιο λοιπόν δεν εκπροσωπεί τα 27 κράτη-μέλη. Μάλλον δεν εκπροσωπούνται στη συζήτηση αυτή τα 27 κράτη-μέλη. Το Κοινοβούλιο συζητά εδώ και πολύ γερό με το Συμβούλιο και την Κομισιόν, εν μέρη σε επιτυχές επίπεδο, για να μπορέσει να καταλήξει ένα οριστικό αποτέλεσμα. Ένα από τους λόγους της δυσκολία είναι ότι δεν μπορούν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι τρίτων κρατών να χωριστούν σε κράτη πρώτης κατηγορίας και δεύτερης κατηγορίας είναι κάτι το οποίο είναι αυτονόητο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν μπορεί ένα κράτος μέλος να θεωρείται πιο σημαντικό ή να έχει μεγαλύτερη αξία από ό,τι αλάκρια από άλλα κράτη-μέλη. Επομένως αυτό είναι σημαντικό σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο επιτρέπουμε σε τρίτια κράτη να αντιμετωπίσουν τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολλές φορές συμφέροντα που πριτανεύουν σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, αλλά δεν μπορούμε εμείς να αλλάξουμε τη μορφή της συζήτησης και να την κάνουμε μια συζήτηση η οποία έχει κατά κάποιο τρόπο εμπορικό χαρακτήρα και ένα χαρακτήρα προτιμήσεων. Θα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να εξασφαλίσουμε ότι εναντί των ΗΠΑ ή του Καναδά υπάρχει μια συνολική ρύθμιση για τα θέματα της αμοιβαιότητας, της προξενικές θεωρήσεις. Επίσης, ένα άλλο ερώτημα είναι το πόσο παίρνουμε στα σοβαρά τις ίδιες τις θέσεις μας. Η Κομισιόν έχει μια θέση η οποία αφήνει πολύ περιθώριο ερμηνείας και αποτελεί και ένα λόγο ανησυχίας για μας. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη μεταξύ των οποίων και η Αυστρία που υποχρέωθηκαν να παραδώσουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις ΗΠΑ σε αστυνομικές ε, βάσεις δεδομένων για προσωπικά στοιχεία υπό την απειλή του ότι δεν θα την χάνουν πια αμοιβαιότητος στις ε, διευκολύνσεις για προξενικές θεωρήσεις. Αυτό η Κομισιόν δεν το έχει διαφυσβητήσει το ότι είναι γεγονός ότι έγινε κάτι τέτοιο. Και υπάρχουν λοιπόν κάποιες χώρες οι οποίες δεν ε, καλύπτονται από μια, επειδή δεν καλύπτονται από μια κοινή στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθενται σε μια τέτοια αμήχανη θέση, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν δημιουργεί ασφάλεια δικαίου και δεν μας βοηθά να έχουμε κάποια ασφάλεια σε σχέση με αυτές τις ε, συμφωνίες. Η Επιτροπή Εξωτερικών απέριψε την πρόταση για αυτά τα θέματα Δυστυχώ με μία μοναχαψήφο διαφορά, θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί το Κοινοβούλιο να καταλήξει σε μία κοινή στάση η οποία να είναι διακομματική για τα θέματα αυτά, για τα μέτρα αυτά τα οποία προβλέπουν μία αμοιβαιότητα για τα θέματα των προξενετικών ε, θεωρήσεων. Είναι λοιπόν σημαντικό το Κοινοβούλιο να μπορέσει να έχει την υποστήριξη της Κομισιόν ώστε να πιέσει το Συμβούλιο να υπάρξει μια κοινή στράχη για τα θέματα αυτά και να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Και ελπίζω ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2013 αυτό θα γίνει πραγματικότητα. Πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία με την Κομισιόν και αν γίνει κάτι τέτοιο δεν μπορώ να φανταστώ το Συμβούλιο να εμποδίσει μια συμφωνία. Ευχαριστώ κύριο Σένσιο. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc Comisiei pentru prezentarea acestui raport. Este al șaptelea an în care acesta se face, dar aș vrea să remarc un singur lucru, că aceste rapoarte, de fapt, descriu numai starea... Για την έβδομη έκθεση αυτού του είδους, αλλά μπορώ να πω ότι αυτές οι εκθέσεις ουσιαστικά δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά μια επισκόπηση της κατάστασης και δυστυχώς δεν περιλαμβάνουν συγκεκριμένες προτάσεις για λήπτεα μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο παραδείγματος χάρη σε θέματα όπως αυτό η αμοιβαιότητα για τις υποξενικές θεωρήσεις. Δεν φταίει φυσικά η Κομισιόν, φταίει η νομοθεσία η οποία υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί εκεί δεν προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα μέσω των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να ασκήσει πίεση για τα κράτη-μέλη επί των κρατών μελών που παραβιάζουν την αρχή της αμοιβαιότητας όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. παραμένουμε σε επίπεδο διπλωματικών διαπραγματεύσεων. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις μέσα αυτό των διαπραγματεύσεων, αλλά αυτό είναι φανερό ότι δεν λειτουργεί. Εγώ υποστηρίζω τη θέση του κυρίου Άλβαρο για τον νέο αυτό μηχανισμό αμοιβαιότητος, του μηχανισμού αυτού λοιπόν ο οποίος έτυχε διαπραγματεύσεων μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου Ελπίζω ότι αν αυτός ο μηχανισμός τελικά γίνει δεκτός οριστικά, θα μπορέσουμε με τον τρόπο αυτό να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και πιο πιστικοί στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα τρίτα, τα τρίτα κράτη και την ανάγκη για τα τρίτα κράτη να εφαρμόσουν πλήρη αμοιβαιότητα για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρία ερωτήματα έχω έναντι της Κομισιόν. Καταρχήν για τον Καναδά. Μετά από τη συζήτηση μετά από τις επαφές και τις συζητήσεις που είχε η Κομισιό με τον Καναδά, υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για να εξευρεθεί κάποια λύση στο πρόβλημα αυτό της απαλλαγή από προξενικές θεωρήσεις. Και εγώ ίδιος πήγα στο Καναδά και μίλησα με τον ε, Υπουργό Μετανάστευσης εκεί, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει σαφήνεια σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα. Δεύτερον, οι Ηνωμένε Πολιτείες. Νομίζω ότι εκεί μπορεί να υπάρχει πράγματι ένα πρόβλημα. Γιατί τα κριτήρια που έχουν στις Πολιτείε Πολιτείες ε, για την μη νόμιμη παράταση της διαμονής δεν μπορούν να επαληθευτούν γιατί δεν λειτουργεί σωστά το σύστημα εισόδων-εξόδων στις ΗΠΑ και έτσι δεν μπορεί να διακριβώσει κανείς ποιοι, πόσα είναι τα άτομα τα οποία έχουν ξεπεράσει την νόμιμη διάρκεια παραμονή του. Τέλος, για την Ιαπωνία δεν έχω καταλάβει τι θα προκύψει μετά την 31η Δεκεμβρίου 2012 όταν η συμφωνία με τη Ρουμανία θα εκπνεύσει. Δεν ξέρω αν θα ε, παραταθεί η ΣΥΣ αυτής της συμφωνίας ή όχι και πού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή. Εγώ κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να χαιρετήσω τις ε, ε, πρόοδους που έχουν επιτευχθεί σε σχέση με τη Βραζιλία, την Ιαπωνία και τον Μπρουνέι. Βλέπω ότι υπάρχουν ακόμα κάποια συνέα. Βλέπω ότι υπάρχουν ακόμα προβλήματα με τον Καναδά. Δεν μας ε, και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρω ότι δεν είναι αυτό εκπληκτικό γιατί είναι χώρες οι οποίες έχουν ιδιαίτερη επιμονή για την πολιτική προξενικών θεωρήσεών τους. Θα ήθελα η Κομισιό να μας πει για το, το, το σύστημα αυτό, ποιες είναι οι προόδοι που προβλέπονται και το χρονοδιάγραμμα μας αναφέρθηκε και στις επιλογές push ή pull, έλξης ή όθησης για τον Καναδά. Ε, πρόκειται για τους, ε, περισσότερο για αυτούς οι οποίοι είναι σε άσυλο και ποιες είναι οι προθέσεις της Κομισιόν για τα θέματα αυτά. Έχουμε ακόμη κάποια σημεία που πρέπει να συζητήσουμε, τα οποία είναι αλληλοσυνδεόμενα. Το σημείο 17 που περιλαμβάνει την έκθεση για τη Συμφωνία ΕΚΑ Ουκρανίας ε, σε σχέση με την έκθεση θεωρήσεων ε, και τη σχέση Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τη Δημοκρατίας του Μόλτοβα για την διευκόλυνση χορήγησης θεωρήσεων. Και για τις δύο αυτές θα έχουμε ε, παρουσιάσει από τον κύριο Ντεκόιστερ, τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Έτσι λοιπόν θα πρότεινα μήπως εσείς ε, να απαντήσετε καταρχήν σε ερωτήσεις, αλλά να προχωρήσετε και στα επόμενα θέματα, γιατί ο κύριος Μουράης ε, είναι αρμόδιος ε, για την Ουκρανία, είναι εισηγητής και ίσως αφού ακούσει την παρουσίασή σας να θέλει να πάρει το λόγο. Παρακαλώ, κύριε Τεκόιστερ. Ευχαριστώ. Φυσικά σήμερα είχαμε την πρώτη παρουσίαση και την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την έκθεση αυτή. Ήδη είμαστε στο 2013. Στο 2013 θα συζητήσουμε όλα τα θέματα που τίθενται στην έκθεση. Έτσι λοιπόν είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα να συνεχίσουμε στην ανταλλαγή απόψεων μαζί σας για το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ερωτήσεις που τέθηκαν. Καταρχήν, για αυτή την ε, συνεργασία για την επιβολή του νόμου, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έπρεπε να προσπαθήσει να συνάψει συμφωνία στο δικό της επίπεδο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να μην ε, ε, περιμένει να συνάψουν διμερείς συμφωνίες στα κράτη-μέλη. Τότε ήταν δύσκολο γιατί τότε είχαμε θέματα τρίτου πυλώνα. Ανήκαν τα θέματα αυτά στο τρίτο πυλώνα και δεν υπήρχε εξωτερική αρμοδιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το τώρα έχει, μάλλον τη στιγμή που καταργήθηκαν οι πινώνες, όλα τα θέματα εμπίπτουν στην εξωτερική αρμοδιότητα, αλλά μέχρι τότε, ε, μέχρι να γίνει αυτή η αλλαγή, τα περισσότερα κράτη-μέλη είχαν δει συνάψει διμερείς συμφωνίες. Ε, τότε ε, θα έπρεπε να είχαμε ζητήσει εντολή για να αντικαταστήσουμε όλες αυτές τις συμφωνίες και θα έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει πιθανότατα πολύ μακροσκελείς διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό θα είχε δώσει ε, την πρόφαση στις Ηνωμένες Πολιτείες να, να βάλει την ένταξη των νέων κρατών μελών στην, στο πρόγραμμα απαλλαγή υποχρέωση θεώρηση. Ακόμη και αν δεν σα αρέσουν δηλαδή οι διμερεί συμφωνίε, υπάρχει μια εξήγηση ιστορικού χαρακτήρα. Και υπάρχουν και λόγοι αποτελεσματικότητα, γιατί πολλά κρατημέλη ήδη είχαν συνάψει τέτοιε συμφωνίε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πιθανό χρονοδιάγραμμα για τον Καναδά και τι ΗΠΑ, για τι ΗΠΑ ε, πολλά θα εξαρτηθούν από την υιοθέτηση νέα νομοθεσία για την απαλλαγή υποχρέωση θεώρηση. Θα δούμε λοιπόν πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα στο Κογκρέσο για τον Καναδά. Όπω είπα στην πρώτη μου παρέμβαση, πιστεύουμε ότι με τη θέση σε ισχύ τη νέα νομοθεσία περί ασύλου. Αυτό θα αποτελέσει αποτρεπτικό. Θα πρέπει να υπάρξει μείωση στον ε, αριθμό των ε, τον ασύλου με ψευδή κίνητρα και έτσι λοιπόν αυτό θα πρέπει να επιτρέψει στον Καναδά να αποφασίσει να την απέτηση θεώρησης τουλάχιστον για τους Τσέχους πολίτες, αλλά και πιθανόν αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για τους Ρουμάνους και Βουλγαρούς πολίτες. Δεν έχουμε λοιπόν κάποια προθεσμία εδώ, αλλά θα δούμε ποιος θα είναι ο δίκτυπος αυτής της νομοθεσίας καταρχήν. Είμαστε σε συνεχείς επαφές με τις καναδικές αρχές για να δώσουμε συνέχιση στο θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά στην Ιαπωνία, ακόμη δεν ε, έχει ληφθεί απόφαση να παραταθεί η προσωρινή απαλλαγή ε, υποχρέωσης θεώρησης για τους Ρουμάνους. Εμείς ε, επιμείναμε να δράσουν κάπως νωρίτερα από τις 28 Δεκεμβρίου που είχαν πει, αλλά τώρα ολοκληρώνουν το σχέδιο απόφασης, όμως δεν θέλουμε να βγούμε εκτός χρονοδιαγράμματος με την Ιαπωνία. Σε ό,τι αφορά το τελευταίο ερώτημα για την ΕΣΤΑ, και τη σχετική έκθεση θα αξιολογήσουμε το σύστημα ΕΣΤΑ αν είναι ισοδύναμο σε διαδικασίες θεώρησης ή όχι όταν εθετηθεί ο τελικός κανόνας γιατί ο τελικός κανόνας μπορεί να επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση και τη σημερινή λειτουργία της ΕΣΤΑ για τις ΗΠΑ προτιμούμε να περιμένουμε. Κατόπιν είχαμε ε, ερώτηση για τους παράγοντες που ε, pull, έλκυσης και όθησης. Ε, πιστεύουμε ότι το σύστημα με τα πολύ ψηλά επιδόματα που ήταν πολύ γενναιόδωρο προσέλκυε ανθρώπους που στην πραγματικότητα δεν έχριζαν διεθνούς προστασίας. Και αυτό έγινε σημαντικό άχθος για τον Καναδά. Από την άλλη, πράγματι υπήρξαν πολίτες των κρατών μελών που ζούσαν σε συνθήκες ε, ανέχειας, ε, ανήκαν σε μειονοτικές ομάδες, δεν τους ε, συμπεριφέρονταν, δεν τους μεταχειρίζονταν σωστά, που ζήτησαν σε κάποιες χώρες όπως ο Καναδάς άσυλο. Σε λίγες περιπτώσεις προσφέρθηκε προστασία και γι' αυτό ο Καναδάς ζητά επίσης να εργαστούμε Επιτροπή των Παραγόντων όφηση στα κράτη-μέλη και να δούμε αν ε, μέσω κάποια μορφή συνεργασία ε, και ανέφερα πριν του χάρη την ορθή ενημέρωση που πρέπει να χορηγηθεί για την νομοθεσία περί ασύλου στον Καναδά. Ε, ζητούν λοιπόν μια τέτοια συνεργασία. Και νομίζω ότι πράγματι υπάρχουν τέτοιοι παράγοντε που σε πουλ. Επομένω, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κομισιόν θα πρέπει να έχουν μια ανοιχτή στάση απέναντι σε μια τέτοια συνεργασία. Όμω, κινδυνεύω να επαναληφθώ, δεν πρέπει να δημιουργηθούν ε, νέες προποθέσει ε, για την ε, άρση τη επαλλαγής υποχρέωση θεώρηση για τα ένα από μήνα τα κράτη-μέλη. Και αν συμφωνείτε πρόεδρε τώρα, να περάσω στα επόμενα δύο σημεία. Θα ήθελα να αναφερθώ από κοινού στην νέα συμφωνία διευκόλυνσης χορήγησης θεώρησης με την Ουκρανία και για τη Μολδαβία Φυσικά πρόκειται για δύο διαφορετικούς φακέλους ε, που θα πρέπει να κρυθούν ανάλογα με τα δικά τους χαρακτηριστικά, όμως δεν θα πρέπει να ε, κρύψουμε ότι υπάρχουν αρκετέ ομοιότητες μεταξύ των δύο αυτών φακέλων. Επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω ότι οι συμφωνίες διευκόλυνση χορήγηση θεώρηση με Ουκρανία και Μολδαβία ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2008 η Κομισιόν έκανε μια αξιολόγηση της λειτουργίας ε, των συμφωνιών διευκόλυνσης χορήγησης θεώρησης το 2009 και επεσήμενε ορισμένες δυσλειτουργίες και δυσκολίες ερμηνείας. Ήδη αυτό αποτελούσε επαρκή βάση για να πούμε ότι υπήρχε ανάγκη αναθεώρησης ε, αυτών των συμφωνιών και θα πρέπει να ευστήσω την προσοχή σας στο ότι αυτή η έκθεση αφορούσε όλες τις συμφωνίες διευκόλυνσης χορήγησης θεώρησης και με πέντε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Φυσικά Μπορώ να σας πω ότι αυτές οι χώρες εν μεταξύ απέκτησαν ε, την ε, απαλλαγή υποχρέωσης θεώρησης. Ε, επομένως, είναι πεπερασμένες οι συμφωνίες και η Κομισιόν τώρα απέκτησε εντολή σε σχέση με τη Ρωσία να επαναδιαπραγματευτεί αυτή τη συμφωνία διευκόλυνσης θεώρησης, αλλά εδώ οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. Γι' αυτό σε αυτό το στάδιο προχωρήσαμε μόνο με τις συμφωνίες ε, τις αναβαθμισμένες για Μολδαβία και Ουκρανία. Και αν σας αναφέρω κάποια νούμερα. Πέρσι στην Ουκρανία είχαμε 1.142.000 αιτήσει θεώρηση. στη Μολδαβία 54.700 αιτήσει Εξετάσαμε αυτές τις συμφωνίες βάσει της λειτουργίας ή δυσλειτουργίας, όπως ε, παρουσιάζεται στην έκθεση αξιολόγησης της Κομισιόν. Επίσης θα θυμάστε ότι οι συμφωνίες αυτές ήταν αντικείμενο διαπραγμάτευσης το 2006-2007. Επομένως, πολύ πριν ε, την υιοθέτηση του κώδικα θεωρήσεων που τροποποίησε εντελώς τις συνερεμονισμένες διαδικασίες χορήγησης θεώρησης και τις προϋποθέσεις. Έτσι, λοιπόν, έπρεπε να προσαρμόσουμε τις συμφωνίες διευκόλυνσης σε αυτή τη νέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ανοίξω μια παρένθεση. Ίσως θα πρέπει να τονίσω ότι σε αντίθεση με τη συμφωνία με τη Ρωσία, οι συμφωνίες με την Μολδαβία και την Ουκρανία δεν ήταν αμοιβές. Δηλαδή οι δικοί μα πολίτε δεν χρειάζονται θεώρηση για να ταξιδέψουν σε αυτές τις δύο χώρε. Γι' αυτό λοιπόν όταν ε, αναθεωρήσαμε τη συμφωνία πρέπει να λάβουμε υπόψη και ορισμένες ε, επιθυμίε που εκφράστηκαν από τι τρίτε χώρε αυτέ. Και νομίζω ότι συνολικά οι, διευκόλ... οι συμφωνίες διευκόλυνσης χορήγησης θεώρησης λειτουργήσαν καλά. Η άρνηση για την Ουκρανία είναι 3,3%. Το ποσοστό άρνησης θεώρηση. Ε, και τη Μολδαβία είναι 9,7, κάπως πιο ψηλό. Όμως, οι πιο σημαντικές διευκολύνσεις που προσφέρονται είναι ότι ε, έχουμε κάποια έκδοση θεώρησης πολλαπλού σκοπού σε κάποιες κατηγορίες πολιτών και για την Ουκρανία έχουμε 35% των θεωρήσεων που εκδίδονται ως πολλαπλών εισόδων και για τη Μολδαβία 23%. Επομένως η συμφωνία για τα σημεία αυτά έχει ήδη λειτουργήσει καλά, όμως ε, φυσικά μια βελτίωση πρέπει να τεθεί κατά νου και διεύρυνση του πεδίου Το κείμενο που έχετε ενωπιόν σα επιφέρει αλλαγέ σε διάφορε πτυχέ. Θα θυμάστε ότι Μία από τις πρώτες διευκολύνσεις αφορά την απλούστευση των συνοδευτικών εγγράφων. Για την Ουκρανία κάποιες νέες κατηγορίες έχουν προσθεθεί στις και φυστάμενες κατηγορίες έχουν διευρυνθεί. Για τη Μολδαβία Κάποιες υφιστάμενες κατηγορίες έχουν διευρυνθεί για οικογενειακές επισκέψεις λόγου χάρη. Δεν έχουμε μόνο τώρα τη διευκόλυνση για τους Ουκρανούς πολίτες που επισκέπτονται μέλη της οικογένειάς τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι Ουκρανοί πολίτες, αλλά αφορά και τους Ουκρανούς πολίτες που θέλουν να επισκεφθούν πολίτες ε, υπηκόους Ευρωπαϊκής Ένωσης, που όμως είναι μέλη της οικογένειάς τους. Αυτό ήταν ένα κενό που έλειπε στην εφτάμενη συμφωνία ένα παραθυράκι. Και επίση οι διατάξει στι θεωρήσει πολλαπλών εισόδων και στι δύο συμφωνίε έγιναν πολύ πιο ακριβεί. Ορισμένε κατηγορίε και οι δύο συμφωνίε τονίζουν ότι οι θεωρήσει πολλαπλών εισόδων πρέπει να εκδίδονται και να ισχύουν μέχρι πέντε έτη. Τι σημαίνει αυτό μέχρι πέντε έτη. Μπορώ να σας πω ότι τα προξενία ε, όταν ε, καθόριζαν το πόσο θα διαρκεί σχέση με αθεώρηση ε, λειτουργούσαν αρκετά αυθαίρετα και δεν είχαμε και τόσες πολλές τέτοιες θεωρήσεις που διαρκούν πέντε έτη. Τώρα, στις διατάξεις η αρχή είναι ότι για τις κατηγορίες τις ενδιαφερόμενες ε, η διάρκεια θα πρέπει να είναι η εγκυρότητα, θα πρέπει να είναι πέντε έτη, εκτός από τις περιπτώσεις που διευκρινίζονται στην ίδια τη συμφωνία. Για την Ουκρανία, το σύστημα του τέλους κατεπήγοντος αναθεωρήθηκε. Ένα τέλος κατεπήγοντος μπορεί να επιβληθεί αν ε, ζει μακριά από το προξενείο ο πολίτης ετών ε, και ζητήσει να διεκπαιρεωθεί αίτησή του σε πολύ σύντομη χρονική περίοδο χωρίς να πρέπει να περιμένει για τις 10 μέρες ε, που προβλέπονται στη συμφωνία. Με τέτοια διάταξη δεν υπάρχει στην συμφωνία με τη Μολδαβία, δεν έχει προσθεθεί. Τώρα, για την άρση του τέλους, ε, καταβολής του τέλους. Ε, έχουμε κάποιες πρόσθετες κατηγορίες στη συμφωνία με την Ουκρανία. Νομίζω μόνο μια κατηγορία για τη Μολδαβία, γιατί ήδη υπήρχε ένας μακρύτερος κατάλογος κατηγοριών που υποφελούνταν ε, από την καταβολή του τέλους από την αρχή. Τώρα, ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι ότι έχουμε προσθέσει διατάξεις και στις δύο συμφωνίες σχετικά με το outsourcing, την υπεργολαβία πάνω κάτω ε, ακολουθήσαμε τις διατάξεις που έχουμε στον κώδικα θεωρήσεων, γιατί στο παρελθόν αυτές οι δύο χώρες είχαν δηλώσει ότι έχουν αμφιβολίες σε σχέση με την ομιμότητα του επιπλέον τέλους που πρέπει να καταβληθεί στην περίπτωση outsourcing, γιατί είπαν ότι η τιμή για τη θεώρηση γενικά τίθεται στη Συμφωνία Διευκόλυσης και είναι 35 ευρώ ενώ αν υπάρχει υπεργολαβία, π.χ. χάρη, αν έχουμε 25 ε, ευρώ παραπάνω που πρέπει να καταβάλλονται ω τέλο υπεργολαβία, αυτό είναι κατά παραβίαση τη συμφωνία. Έτσι λοιπόν τώρα προσθέσαμε τις κατάλληλε διατάξεις για το outsourcing, την εξωτερική ανάθεση. Και τώρα φτάνω στο τελευταίο σημείο, γιατί είναι και πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε την άρση απαλλαγή για τα περισσιακά διαβατήρια. Στι τέτοιε συμφωνίε ε, ήδη ίσχυε κάτι τέτοιο για τα διπλωματικά διαβατήρια, του κατόχου διπλωματικών διαβατηρίων από Μολδαβία και Ουκρανία. Νομίζω ότι είναι μια κανονική εξέλιξη το πεδίο εφαρμογή ε, αυτή τη απαλλαγή να διευρυνθεί και πράγματι τα κράτη-μέλη υιοθέτησαν μια τέτοια απαλλαγή για τα υπηρεσιακά διαβατήρια, για τους κατόχους του στην περίπτωση που είναι βιομετρικά. Και εδώ να προσθέσω ότι για την Ουκρανία τα υπηρεσιακά διαβατήρια δεν είναι ακόμη βιομετρικά. Στη Μολδαβία είναι. Όμως προσθέθηκε μια δήλωση για την Ουκρανία ότι φυσικά αν υπάρξει κατάχρηση αυτής της απαλλαγής υποχρέωσης θεώρησης ή αν προκύψουν προβλήματα δημόσιας τάξης, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αναστείλει την εφαρμογή της διάταξη αυτής. Με τη Μολδαβία το ίδιο κείμενο έχει τεθεί επί χάρτου και το κείμενο έχει εγκριθεί από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτή τη στιγμή η Κομισιόν παρουσίασε τις αποφάσεις ε, και Υπήρξαν κάποια αρνητικά σχόλια για αυτή την απαλλαγή υποχρέωση θεώρηση ε, για του κατόχου υπηρεσιακών διαβατηρίων τη Ουκρανία. Υπόθηκε ότι δεν ήταν καλή ιδέα, λαμβάνοντα υπόψη τι ε, συνολικέ σχέσει με την Ουκρανία και την κατάσταση σε σχέση με το κράτο δικαίου κτλ. Αλλά ο Επιτροπό μα ε, δήλωσε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και άλλοι εκπρόσωποι τη Κομισιόν στην ΑΦΕΤ, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, να συζητήθηκε το θέμα, ότι με την πρόβλεψη νέων κατηγοριών όπως εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και συγκεκριμένες διευκολύνσεις για νέους κτλ. Αυτό δεν ε, ήταν δώρο προς την κυβέρνηση αυτή η συμφωνία, αλλά δώρο προς ε, τον πληθυσμό της Ουκρανίας, τον Ουκρανικό λαό. Έτσι λοιπόν το ότι υπάρχει αυτή η απαλλαγή υποχρέωσης θεώρησης για τους κατόχους υπερσιακών διαβατηρίων δεν θα πρέπει να αποτελεί λόγο να μπλοκαριστεί η κύρωση. Πρόεδρε, αυτή είναι η επισκόπηση των πιο σημαντικών στοιχείων ε, ε, των αναβαθμισμένων συμφωνιών με Μολδαβία και Ουκρανία. Έχουν υπογραφεί 23 ε, Ιουλίου και 27 Ιουνίου αντίστοιχα. Επίσης ξέρετε ότι με αυτές τις δύο χώρες ο διάλογος απελευθέρωσης που συνεχίζεται. Αυτές οι ε, νέες συμφωνίες θα πρέπει να θεωρηθούν ως ένα επόμενο βήμα προς τον τελικό στόχο. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ κύριε Ντεκόστερ. Μετά από αυτή την παρουσίαση της Κομισιόν, την συνοπτική παρουσίαση της Κομισιόν, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μωράης, ο οποίος είναι εισηγητής για τα θέματα της Ουκρανίας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξέρω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Και γι' αυτό θα, απαντήσω, θα προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτά που είπε η Θα προσπαθήσω να έρθω στην ουσία. Από την παρουσίαση της Κομισιόν μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι υπήρξαν κάποιες τεχνικές προσαρμογές στη Συμφωνία που αποτελούν πραγματική βελτίωση για τους πολίτες της Ουκρανίας. Από την πλευρά μας του Κοινοβουλίου πιστεύω ότι υπάρχει ένα πολιτικό στοιχείο. Την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια συζητήσαμε την κατάσταση στην Ουκρανία στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων που είναι η κύρια επί της ουσίας επιτροπή, φυσικά και εμείς εμπλεκόμεθα και η Κομισιόν και συζητήσαμε για τα συστήματα αυτά προξενικών θεωρήσεων δεν πρέπει να ανταμείψουν την κυβέρνηση της Ουκρανίας αλλά αντίθετα το λαό της Ουκρανίας. Η δική μου άποψη είναι ότι εάν δείτε το ποσοστό απόρριψης που είναι 3,3% το γεγονός ότι το σύστημα αυτό λειτουργήσε καλά τότε οι προτάσει κομισιών, η κατάργηση του τέλους ε, προξενικής θεώρησης που είναι 70 ευρώ, οι προξερικές θεωρήσεις πολλαπλής ε, εισόδου, η ε, κατάργηση της υποχρέωσης βίζας για σύντομη αμονή, όλα αυτά είναι θετικά στοιχεία που θα δώσουν περισσότερες δυνατότητε στους πολίτες Ουκρανίας με τη συμφωνία αυτή, αλλά μετά και τη συζήτηση μέσα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων υπάρχει και ένα πολιτικό θέμα. Από τη δική μας πλευρά θεωρώ ότι είναι μια καλή συμφωνία και οι τροποποίησεις της Κομισιόν είναι πολύ θετικέ και εγώ τις υποστηρίζω πλήρως έχοντας παρακολουθήσει όλο αυτό το θέμα Μπορώ να πω λοιπόν ότι είμαι ικανοποιημένο με αυτά τα οποία έχουν συμβεί, αλλά δεν πρέπει να λησμονήσουμε την πολιτική διάσταση και να τονίσουμε ότι έχουμε ένα πολιτικό εργαλείο το οποίο έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε μέσα σε μια πολύπλοκη κατάσταση. Η ΑΦΕΤ θα αποφασίσει στις 22 νομίζω Ιανουαρίου και αυτό μπορεί να αλλάξει φυσικά ως ημερομηνία, αλλά για σήμερα εγώ θα ήθελα να ακούσω απόψεις, εάν υπάρχουν απόψεις, από τους λίγους και εκλεκτούς συναδελφούς που έχουν μείνει. Και κάνει και κρύο εδώ κύριε Πρόεδρε. Μόνο εγώ κρυώνω ή κρυώνουν και άλλοι. Εγώ έχω τουρτουρίσει εδώ. Επειδή έρχομαι από το Ηνωμένο Βασίλειο με εκπλήσει αυτό. Εν πάση περιπτώσει έχουμε αναμείνει την Ουκρανία ένα μεγάλο διάστημα για να υπάρξει αυτή η συμφωνία. Περιμένουμε λοιπόν για την ψηφοφορία στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Αν υπάρχουν όμω κάποιε απόψει για αυτό το θέμα, μετά και από τη συζήτηση τη Ολομέλεια, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω τι απόψει συναδέλφων που ενδεχομένω έχουν μεγαλύτερη εμπειρία για τα θέματα αυτά. Βάσει της διαδικασίας όμως, νομίζω ότι είναι πολύ καλές αυτές οι τροποποίησεις και θα παρακολουθήσω φυσικά και τη διαμόρφωση απόψεων στην ΑΦΕΤ. Ευχαριστούμε κύριε Μωράης. Δεν πρέπει να θέλετε υπερβολικό βάρος στους ώμους σας. Θα έρθει ο Άγιος Βασίλης και θα βοηθήσει. Δεν ξέρω αν είναι πιο ζεστά όμως στις άλλες επιτροπές και στον, διάλογο τριγωνικό διάλογο από την εδώ πέρα. Μην ανησυχείτε, λέει ο πρόεδρος. Ο κύριος Προτάσιεβιτς έχει να προτείνει κάτι. Το ίδιο αισθάνεστε, κρυώνετε κι εσείς. Ο κύριο Προτασίεβιτς, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μιλήσω πολωνικά. Σύντομα, ξέρω ότι δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μας προβληματιζόμαστε όχι μόνο για θέματα ασφαλείας και πολιτικών ελευθεριών εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά εξετάζουμε και την κατεύθυνση προς την οποία να αλλάζουν τα πράγματα στη γειτονιά μας. Και από αυτή την άποψη ε, θα ήθελα να θεωρήσω να εξετάσω το θέμα αυτό της διευκόλυνσης ε, του καθεστώτος θεωρήσεων ε, προξενικών για την Ουκρανία. Είναι μια θετική αλλαγή που θα λάβει η χώρα. Κάτι που θα επηρεάσει και πολλούς Ουκρανούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από τη σύγκριση των δραστηριοτήτων των πολιτών. Δραστηριοτήτων που, στη, που, έχουν, μπορούν να ασκήσουν στη χώρα τους και στις χώρες. Κυρίως χώρες που ξεκίνησαν από παρόμοια θέση κατ' παρελθόν και έφτασαν σε σημερινή κατάσταση, όπως η Πολωνία, η Τσεχία και οι Βαλτικές χώρες. πολίτες, δημοσιογράφοι και μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων και θρησκευτικών ομάδων που συμμετέχουν στις ανταλλαγές μεταξύ χωρών, φοιτητές, και διάφοροι άλλοι κάνουν αυτές τις συγκρίσεις. Ξέρουμε από έρευνες ότι οι Ουκρανοί που έχουν πάει σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης περιμένουν θετικές αλλαγές να λάβουν χώρα και στη χώρα τους και να πλησιάσει η χώρα τους τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η συμφωνία που παρουσιάστηκε εκτενώς και λεπτομερώς από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τεχνικές πτυχές αλλά και πολιτικές και πολιτικό βάρος. Και όσο πιο σύντομα γνωμοδοτήσουμε θετικά εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τόσο το καλύτερο για τις μελλοντικέ μας σχέσεις με τη σημαντικότατη αυτή γειτονική χώρα που κατέχει και στρατηγική θέση στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχουν άλλες ε, παρεμβάσεις και δεν βλέπω να έχουν σηκωθεί άλλα χέρια, στρεφόμαστε και πάλι στον κύριο Τεκλόιστερ για να ολοκληρώσει το θέμα αν θέλει να πει κάτι από πλευρά τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν είστε υποχρεωμένο, αν δεν θέλετε, εντάξει. Οπότε τελειώσαμε για την ώρα. Ευχαριστώ για τη συζήτηση. Ακριβώ την ώρα μα. και θα ακολουθήσει η συνεδρία των συντονιστών που θα λάβει χώρα σε μερικά λεπτά. Ετοιμαζόμαστε για τη συνεδρία και των θύρων και ελπίζουμε να υπάρξουν αρκετοί συντονιστές για απαρτία για να λάβει χώρα η συνεδρία των συντονιστών. Ευχαριστώ.